Ναι. Buonasera, inizio i lavori di questa commissione. Καλησπέρα σας. Αρχίζουν οι εργασίες της Επιτροπής μας. Τι Έχουμε καταρχήν την υιοθέτηση της έκθεσης Ντουργκάης για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της ε, σύνδεσης Λιών το Ρήνο με το τρένο μεγάλης ταχύτητας ε, Επίσης, αποστολή στην Βουλγαρία και σχετική έκθεση, ε, συνάντηση με τον Πολωνό, με την Πολωνή ε, διαμεσολαβήτρια, την κυρία Ειρήνη Μιλκόβιτ και έπειτα έχουμε και το θέμα των διακρίσεων φίλου και την ε, ομοφοβία. Ρωμανία, ένα θέμα το οποίο έχουν υποβάλει ε, ετούμενοι από διάφορες χώρες. Ζητώ από του συναδέλφου να εγκρίνουν την ημερήσια διάταξη. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται η σημερινή ημερήσια διάταξη. Σα θυμίζω ότι η... έχουμε τρει συνεδρίαση τρει μισέ ημέρε και την πέμπτη έξι του μηνό θα γίνει το σεμινάριο που έχουμε διοργανώσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι θα υπάρξει μαζική παρουσία την ημέρα του σεμιναρίου από πλευρά των συναδέλφων, κυρίω στο πρωινή σύνοδο τη Επιτροπή μα. Να θυμίσω εξάλλου ότι η Πολωνή διαμεσολαβήτρια, η καθηγήτρια Λιπόβιτσε θα υποβάλει δήλωση αύριο το πρωί στη Κομισιόν, ενώ θα πρέπει να εξεταστούν και ε, αναφορές οι οποίες ε, προέρχονται από την Πολωνία. Όσον αφορά την αναφορά 1557 του 2009, που προβλέπεται να εξεταστεί στην ημερήσια διάταξη στο σημείο 10 έχει μεταφερθεί μετά από αίτημα των αναφερόντων και της συναδέλφου Άνκης. Θα είναι παρόντες στην αίθουσα διάφοροι ε, αναφέροντες για τις αναφορές που αναφέρω μόνο με τον αριθμό που είναι γεγραμμένες 6, 7, 9, 15, 17, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 και 32. Πρέπει να εγκριθούν τα πρακτικά της 8 η Σεπτεμβρίου 2011. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά ε, θεωρούμε πως εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Και στο σημείο 3, ως ήθιστε, να σας ανακοινώσω ότι έχουν διανεμηθεί τα παρατήματα και οι συνάδελφοι καλούνται να διαβιβάσουν τις ε, παρατηρήσεις τους για τα παρατήματα Συγκεκριμένα σας ε, σημειώνω την απάντηση που στείλαμε στον κύριο Τεγκεπάουερ μετά από την απόφαση του 10 για την ε, υπόθεση που κατετέθη από τον ε, αναφέροντα αυτόν. Εάν δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, θα περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Στο 5 έχουμε την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων βάσει των αναφορών που ελήφθησαν. Η συγκητής είναι ο συνάδελφος Ιτρουγκάης, στον οποίο θα δώσω το λόγο πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους. Απλώς να ευχαριστήσω όπως ήδη έχω πράξει για την συνεργασία την ε, γραμματεία μας αλλά και όλες τις πολιτικές ομάδες σε σχέση με την έκθεσή μου. Και τέλος πάντων πριν την ψηφοφορία εάν κάτι θα ήθελα να προσθέσω θα είναι η έκπληξη. Ε, Όπω ξέρετε είμαι ο εισηγητής, ο συντάκτης έκθεσης. Την έκ, έλεγα την έκπληξη την οποία ένιωσα διότι τις τελευταίες μέρες της περισμένης εβδομάδα λάβαμε γνώση στο λίγο Κόμμα ότι μία συνάδελφος υπέβαλε σειρά τροπολογιών. Και όπως ξέρετε και θα θυμάστε, ευθύς εξ αρχής εγώ είχα τεθεί στη διάθεση όλων των πολιτικών ομάδων, ούτως ώστε όποτε θέλουν να συναντηθούμε και το είπαμε αυτό έγινε τρεις φορές με τους σκιώδες ηγητές και τους, ε, τους ενημέρωσα και όπως σας έλεγα υπήρξε έκκληση, μια που κόντρα σε κάθε παράδοση, όχι της Επιτροπής, αλλά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, συναντήθηκε με άλλα πολιτικά κόμματα, κρυφά από μένα, ούτω ώστε να υποβάλει, αφού συζητήσει τις τροπολογίες της. Αυτό είναι κόντρα σε κάθε τύπο, σε κάθε ουσία, σε κάθε πρωτόκολλο. Και ξέρουμε ποια είναι είναι σοσιαλίστρια. Η κυρία Μέρκης έπραξε τα αυτά. Και δεν σας το λέω με κακία, με πικρία. Εμείς και εκείνη τη θέλουμε στο πλευρό μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι όσον αφορά τις τροπολογίες της. Επαναλαμβάνω. Δεν λέω ότι θα πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση που μου είναι δυσάρεστη. Αλλά θα πρέπει να μην αφήνουμε περιθώρια να έχουμε τέτοιες συμπεριφορές διασπαστικές όταν υπάρχει δρομολογημένη μια έκθεση σε αυτήν την περίπτωση ήταν η έκθεση του Λεκού Κόμματος. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε αυτό, να μην αποτελέσει προηγούμενο πρόεδρε και να μην έχουμε τέτοιου είδου ατμόσφαιρα σε σχέση τη ε, συνήθου καλή ατμόσφαιρα που έχουμε πάντα σε συνεργασία με σοσιαλιστέ φυσικά, με κύριο Άουκεντο, του πράσινου, με την ε, Νοτική Αριστερά, με τους ε, μη εγγεγραμμένους, με τον κύριο Σαλαβράκο, με όλου, με όλους υπάρχει καλή ατμόσφαιρα, καλό κλίμα. Γιατί όπως σας είπα, όλες οι πολιτικές ομάδες και η γραμματεία, όλοι όλοι, επανειλημμένα, Θέλουμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο άνταρτο πόλεμο και εγκρυπτό και παραδείστο να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε συνάδελφα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που κάνατε. Να ευχαριστήσω και εγώ την γραμματεία και αρχίζουμε την ψηφοφορία. Όχι, η συνάδελφος Όκεν. Να σας πω στα δανέζικα. Ε, ναι, στα δανέζικα. Αγαπητή Πρόεδρε, έχω τα εξή δύο να σα αναφέρω όσον αφορά τα όσα μα είπε και ο πρωτα Πρώτα-πρώτα, ότι θα πρέπει να τον ευχαριστήσω διότι ήταν αγαστή, ήταν θετική, ευχάριστη η συνεργασία μας για την εκθεσή του. πάντω, δεν συμφωνώ 100% σε σχέση με το τι συνέβη και δεν συνέβη. Ναι, ε, ε, έχουμε καθέσει έχουμε κάποιες ρυθμίσεις, κάποιες συμφωνίες και αυτό Μπορώ να πούμε ότι έχει ξαναγίνει, έχει ξαναγίνει μεταξύ σκιωδών και κυρίου εισηγητού. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να δουλεύουμε ακριβώς όπως τα είπατε κύριε. Όμως θα πρέπει και εσείς να συνεχίσετε να ενεργείτε αντικανονικά όπως έχει ήδη γίνει στο παρελθόν. Όχι, ξέρω, δεν έγιναν όλα ρόδινα, αλλά Εντάξει. Ό,τι έγινε έγινε. Θα πρέπει επομένω. Ό,τι έγινε έγινε και από τώρα και στο εξή να γίνουν τα πράγματα όπω πρέπει και πάλι σα ευχαριστούμε συγκητά. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να περιορίσω τη συζήτηση. Ωστόσο, συνάδελφοι, σα παρακαλώ να καταλάβετε ότι ψηφίζουμε τώρα. Ο συνάδελφο που στην ώρα ζήτησε το λόγο, αλλά μόνο ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Τέσσερα. Ε, άκουσαν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος Φιτουργκάης. Ε, ε, όμως κοιτάξτε, για αυτή την πολεμική έχω να πω ότι εδώ πέρα δεν είναι παρούσα η, εν λόγω συνάδελφος. Επομένως δεν είναι πάρα πολύ σωστό τώρα να συζητούμε σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν. Θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα συνεργασίας, εμπιστοσύνης, θα πρέπει αυτό το κλίμα να κατησχύει. Ό,τι περιστάσεις και, και να υπάρχουν, ό,τι και να κάνουμε εδώ στην Επιτροπή Αναφόρων. Ούτε εγώ θέλω να επισελθώ στην ουσία. Ούτε θέλω να αρχίσουμε τώρα κουβέντα, αλλά θέλω να απαντήσω στον συνάδελφο και φίλο Μποστινάρου. Είναι σοβαρό αυτό το περιστατικό. Αν υπάρχει μια συνάδελφο αυτό το οποίο θέλει να κατεβάσει κάποιε τροπολογίε, θα πρέπει να έρχεται σε συνεννόηση με τι άλλε ομάδε. Αλλά θα πρέπει να το λέει και στον εισηγητή. Τι λέει, κατεβάζει οι δύο ονόματι τροπολογίε και σήμερα δεν εμφανίζεται να ψηφίσει. Μα γιατί το κάνει αυτό, γιατί να γίνονται έτσι τα πράγματα, γιατί δεν μα ειδοποίησε. Σα είπα. Το, το, το, το είπαμε, καλέσαμε οποιονδήποτε θέλει. Είμαστε ανοιχτοί δεν υπάρχει κάτι το οποίο αξίζει να αποκριθεί εδώ. Κοιτάξτε, εγώ συμμερίζομαι την ανάγκη να το συζητήσουμε, όπως είπε και ο, κύριος, ο συνάδελφος Μπουστινάρο, αλλά κάποια άλλη στιγμή. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 38, παράγραφος 1 της συναδέλφου Μέρκης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 στην παράγραφο 1α νέο τη συναδέλφου Αλφάνο σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Σας παρακαλώ να ξανακάνουμε την ψηφοφορία γιατί δεν είναι ξεκάθαρο και πρέπει να μετρήσουμε. Ποιοι είναι υπέρ. πέρα. Euh, Prima parte dell'emendamento, seconda parte 39. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 39. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εμενταμέντο 40 al παράγραφο 2 della collega 40 για την παράγραφο 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 τη συναδέλφου Μέρκη. σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 42, ματσόνι, στην παράγραφο 4, ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Emendamento 44 al κολέγα στο παράγραφο. 44 του συναδέλφου Iturgais ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 της συναδέλφου Μέρκης ε, στην παράγραφο 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 45 ματσόνες στην παράγραφο 6 ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Τροπολογία 46, Μέρκη στην παραγραφή 6, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47, στην παράγραφο 7 της συναδέλφου Μέρκης, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία Κρουγκάη στην παράγραφο 8, η τροπολογία 48, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία Μέρκης 49, στο παράγραφο 9, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία Βάλεαν 51, ε, αφορά την παράγραφο 10α, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50, έχει καταπέσει, 52, Μπουλάντ, στην παράγραφο 11. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 μέρκη στην παράγραφο 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 54 Μέρκης στην παράγραφο 13α. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 55, πάξας, στην παράγραφο 14, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Βάλεαν 56, παράγραφο 14, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57, Μέρκης, παράγραφος 14, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 58, μπουλάντ, παράγραφο 16, α, ποιοι είναι υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 59, Βαλεάν, παράγραφος 18α, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60, Μέρκη, στην παράγραφο 20, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 61, Βάλεαν, στην παράγραφο 25α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62, η Τουργκάη, στην παράγραφο 27, ποιον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 64, Βάλεαν, στην παράγραφο 27α, ποιον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 65, Πάξες, στην παράγραφο 28α, ποιον υπέρ, κατά εποχές απορρίπτεται συμβιβαστική α στην παράγραφο 29 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στην τροπολογία 68 μέρικες. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 69, Μπουλάν, στην παράγραφο 30, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, Ντεμπρούν, στο εκτιμώντας α, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, Μέρκης, εκτιμώντας γ, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4, Μέρκης, στο εκτιμώντα ε, ε, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5, Μέρκης, στο σίγμα ταφ, εφ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6, Βάλεν, στο εκτιμώντας ζήτα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 Αλφάνο, ποιν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 Βαλέντες, εκτιμώντας ε, ε, Ήτα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 Ντεμπρούν στο Ι, ποιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 όκεν στο εκτιμώντας για τα α, κάπα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β στο εκτιμώντα για β, ποιοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 όκεν, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 Μέρκης ε, υπέρ κατά αποχές γκρίνα, ε, απορρίπτεται, με συγχωρείτε. 16 Βαλεάνα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογίες 16 και 10, 17 ε, και 18, και Αλφάνο, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 19 στο εκτιμώντας ταφ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 μπουλάντε το εκτιμώντα ΚΒΒ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 21 ματσόνι ποιοι είναι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 22 μπουλάντε, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 ματσόνι ποιοι είναι υπέρ κατά κα, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία ταυτόσημη ματσόνι Α, συγγνώμη, έκανα λάθο. Τροπολογία 24 ματσόνι. Ποιοι είναι υπέρ, 24. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25, όκεν στο ίδιο εκτιμώντας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 26, ματζόνι, υπέρ, κατά, αποχές. Τροπολογία 27, ματζόνι, ποιοι είναι υπέρ, κατά, από αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 ντεμπρούν, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 μέρκης, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Προφορική τροπολογία. Θέλετε να μας το αναλύσετε. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 30 όκεν όπως έχει τροποποιηθεί. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 31 μπουλάν. Στο εκτιμών... Ε, ε, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 η Τουργκάιθ, Όκεν. Δεμπρούν, Ματσόνι και 32 Δεμπρούν είναι ταυτόσιμες υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογίες 34-35 είναι ταυτόσιμες τις ψηφίζουμε από κοινού ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Τροπολογία 36 Βάλεαν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 37 Ετουρκάις Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 1 Αλφάνο. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνονται. Και τώρα ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον συνάδελφο Ιτουρκάης.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 Λίγη ησυχία. Έχουμε την αναφορά 1.24 του κυρίου Ντάν Πέσκο, του Βρετανού, εξ τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών, του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών, σχετικά με την πρόσβαση των τυφλών στα βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα. Θα δώσω το λόγο για πέντε λεφτά στον αναφέροντα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μέλη της Επιτροπής, αξιότιμοι και κύριοι Ευρωβουλευτές. Ονομάζομαι Christopher Friend. Είμαι τυφλός πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και μιλώ σήμερα υπό την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών και της σχετικής παγκόσμιας εκστρατείας για το τέλος της, ε, ε, της δίψαση για βιβλία. Έχουμε εμπειρίε σε τέτοιου τύπου καθημερινά. Είμαστε καταδικασμένοι σε λογοτεχνική και πολιτισμική ε, ένδια, διότι οι εκδότες που έχουν τα δικαιώματα σε αυτή την περίπτωση δεν παράγουν και δεν διανέμουν ε, το 95% το 95% καλά ακούσατε όλων των έργων που δημοσιεύουν σε μορφή αναγνώσιμη για μας. Κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, σας καλώ να φανταστείτε για μια στιγμή πως ε, αργότερα την ίδια αυτή τη βδομάδα θα πάτε στην τοπική σας δημόσια βιβλιοθήκη και εντός αυτής θα βρείτε ότι το 95% όλων των βιβλίων είναι αλυσοδεμένα και κλειδωμένα και δεν μπορείτε να τα διαβάσετε. Πώς θα αισθανόσασταν εσείς, απογοητευμένοι, θυμωμένοι, θα αισθανόσασταν θύματα διάκρισης, Πάντω σίγουρα εμεί είμαστε δικαιολογημένα πολύ απογοητευμένοι. Εμεί θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία που έχετε κι εσεί να μπορούμε να περπατήσουμε στο κεντρικό δρόμο τη πόλη μα και να μπούμε σε μια δημόσια βιβλιοθήκη, σε ένα βιβλιοπωλείο, ώστε να δανειστούμε ή να αγοράσουμε το τελευταίο best seller με ένα βιβλίο που όλη μας η οικογένεια και όλοι στην πόλη έχουν διαβάσει και το συζητούν τα κράτη-μέλη της WIPO, ε, που είναι ο Διεθνής Οργανισμός για την ε, Πνευματική Διοκτησία, διαπραγματεύονται ένα διεθνές μέσο για τα πνευματικά δικαιώματα που θα αποτελέσει βασικό κομμάτι ε, της ενδεχόμενης λύσης του προβλήματος των βιβλίων. Αυτή η λύση προτάθηκε καταρχήν πριν από 27 ολόκληρα χρόνια σε μια έκθεση που από κοινού είχε, ανατεθεί η WIPO, είχε αναθέσει η WIPO και η UNESCO. Τον Μάιο του 2011 το Ευρωκοινοβούλιο μέσω των, του άρθρου 70 της έκθεσης ε, του Κοινοβουλίου, ξεκλειδώνοντας το δυναμικό της ε, πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, επισήμως κάλεσε την ε, διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην WIPO, δηλαδή τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή, να στηρίξουν μια συνθήκη για, τους, για τα άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν. Είμαι σήμερα λοιπόν εδώ για να σας αναφέρω πως η διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ακολουθούν το κάλεσμα του Κοινοβουλίου. Και μόλις στις 23 Αυγούστου τόσο πρόσφατα ο ίδιος ο Επίτροπος Μπαρνιέ έγραψε εις ένα α, ε, βουλευτή απαντώντας του και ένσα να σας πω ακριβώς τι, τι είπε χρησιμοποιώντα τη μετάφραση του πρωτότυπου του γαλλικού, είπε επιλέξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να ευνοούν ή μάλλον συγγνώμη, συνεχίζουν να τιμούν αυτήν την σύσταση, να την τηρούν. Και μας είπαν ότι υπάρχει αυτή η δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου ε, σύσταση, η οποία μας είπαν ότι είναι πιο ευέλικτη, πιο αποτελεσματική από ό,τι συνθήκη, όμως στην ίδια εκείνη συνάντηση οι διαπραγματευτέ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού ερνήθησαν να μιλήσουν για το τι προβλέπει η συνθήκη για τους τυφλούς με ενθουσιασμό υπεστήριξαν την πρόταση για μια ευρεία διπλωματική διάσκεψη ούτω ώστε να τηρηθεί η συνθήκη για τα οπτικοακουστικά. Και Πρόκειται για κάτι το οποίο το απαιτούν οι δικαιούχοι και είναι αυτό το οποίο γίνεται. Οπότε κάποιο δικαιούχο επικαλείται κάποια σύσταση για να προστατεύσει συμφωνητά του. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει ε, τα δικαιώματα των τυφλών ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Και επίση να αναλάβει τι ευθύνε ε, που προβλέπει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ταυτόχρονα η σύμβαση του ΟΗΕ για τους ε, αναπήρους. Madam Chair, over 100... Κύριε Πρόεδρε, πάνω από 100, 100 του φορέα μας είναι υπέρ ε, του να τηρηθεί συνδίκη όσον αφορά τους τυφλούς και η ΒΑΕΠΟ εάν βοηθήσει και συνθήκη θα μπορούσε να ολοκληρώσει ε, την ε, σχετική μελέτη, τη σχετική συνθήκη μέχρι το τέλος του 2012. Οπότε αυτή, αυτός ο φορέας για τους ε, τυφλούς παγκόσμιος φορέας, ο ευρωπαϊκός φορέας, αλλά και οι συναδελφοί από τον φορέα των δυσλεκτικών αναγνωρίζουν ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στη τελευταία συνεδρίαση ε, copyright του, της WIPO. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη της WIPO ε, τελικά κατάφεραν να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία σε σχέση με ενιαίο κείμενο το οποίο τελικά θα μπορούσε να αποτελέσει κείμενο νόμου. Εάν δε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λάβει τις ευθύνες της τελικά, ούτω ώστε να μπορέσουν οι ανάπηροι να έχουν ε, κάποιο είδους ε, λύση ε, να σταματήσει αυτή η έλλειψη αυτό το, το έλλειμμα όσον αφορά το διάβασμα και τα βιβλία έστω και με δευτερογενές δίκαιο έστω και με ε, ενδοτικού δικαιοδιοτάξης θα πρέπει εμείς κάτι να κάνουμε, θα πρέπει εσείς να, να συντάξετε μια, ένα, ψήφισμα το οποίο να κατέβει προς ψήφιση στην επόμενη ολομέλεια του Κοινοβουλίου σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. παρουσιαστε αυτή την αναφορά. Και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, στην εκπρόσωπο μα θα δώσω πρώτο το λόγο στον κύριο Μακένι από την DG Mark. Σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε, λίγο προς Επιτροπής. Επίσης σας ευχαριστούμε που ακούτε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σήμερα και θα αρχίσω τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρω δεσμευτεί όσον αφορά κάποιες προσπάθειες για να βοηθήσει ε, αυτό το, το, το έλλειμμα, ε, το πρόβλημα, τη φτώχεια σε σχέση με το διάβασμα που είπε ο αναφερόμενος. Και εμεί προσπαθούμε να βρεθεί μια λύση εντός και εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, στα πλαίσια Ευρωπαϊκή Ένωσης έχουμε αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλειών σημαντικών και εδώ θα πρέπει να σταθώ στις ε, πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αμεσότερα σχέση με αυτά τα οποία είπε ο αναφέρον προηγουμένως όσον αφορά το copyright. Βέβαια, έχουν καταβληθεί και άλλες προσπάθειες, έχουν αληφθεί και άλλες προσπάθειες από την Κομισιόν και από ε, άλλε γενικέ διευθύνσει, όπω η Γενική Διεύθυνση για τα θέματα δικαιοσύνη. Δεν θα σταθώ εκεί. Όμω, αν σα ενδιαφέρει, όταν έχουμε ρωταπαντήσει, θα σα πω. Πάντω, έχουμε πρώτα-πρώτα αυτό το copyright, που έχουν πρώτα το θέμα το οποίο απασχόλησε τώρα τον αναφέροντα. Εμείς ξέρετε ήδη έχουμε θεσπίσει νομοθεσία στο επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί ορίζεται ότι έχουν την πιθανότητα τα κρατημέλη, τη δυνατότητα να περιορίσουν τα δικαιώματα ε, των δικαιούχων υπέρ των αναπήρων συμπεριλαμβανομένων και των τυφλών. Και επίσης Πάρα κράτη-μέλη επομένω έχουν ασπαστεί ε, τα σχετικά. Επίσης εμείς βοηθούμε να ε, υπάρχει ε, ευχερής ανταλλαγή βιβλίων σε φόρμα σε μορφή που να είναι προσβάσιμη εύκολα για όλα αυτά για να βοηθήσουμε τους τυφλούς και σε συνεννόηση και με το σχετικό εμπορικό κλάδο και υπογράψαμε ε, ένα σχετικό μνημόνιο ή υπόμνημα ακριβώς για υπέρ των ε, τυφλών το Σεπτέμβριο του 2009 αυτό τον έλαβε ο Επίτροπος Μπαρνιέ και το προσυπέραψαν εκπρόσωποι της, ε, του Φορέα των Τυφλών και του, του, Φορέα των Δυσλεκτικών. Ακριβώς οι φορείς που σήμερα παρέσανται στην αίθουσα αυτή και επίσης παρέστησαν και εκπρόσωποι εκδοτών, συγγραφέων κλπ. Έκτοτε εμείς επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με όλους αυτούς τους εμπλεκομένους, αυτούς όσους θέλησαν να συνεργαστούν μαζί μας, ε, πασχίζουμε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις πρακτικές, εφαρμοστικές λεπτομέρειε αυτού του υπομνήματος, ε, να λάβουμε υπόψη τους πυρισμούς των κρατών μελών και να δούμε πώς θα στήσουμε ένα δίκτυο για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των βιβλίων που θα πρέπει να έχουν ε, στη βιβλιοθήκη τους οι τυφλοί ε, ανταλλαγή των βιβλίων υπό τέτοια μορφή, φόρματα ας πούμε, που να είναι προσβάσιμα σε αυτούς. Τώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόεδρε, ε, όσον αφορά τις εξωτερικές μας δράσεις και εμείς επίσης ε, μπορούμε να αναπτύσσουμε δράση όσο γίνεται πιο έντονα όσον αφορά τις συζητήσεις στην WIPO ε, και προσπαθούμε να βρούμε να γίνει κάποιο είδου διεθνή συμφωνία, να βοηθήσουμε αυτά τα προνεφερθέντα άτομα. Και όπως γνωρίζετε, αυτά τα οποία προσβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια θέση ε, που τα σπάζονται σε συντονισμό μαζί μας και τα κρατη Πρόκειται για θέματα κοινή αρμοδιότητας εθνική και κοινοτική, όπου βέβαια για να αναλάβουμε εμεί δικαίωμα πρωτοβουλία θα πρέπει να πάρουμε εντολή από το Συμβούλιο για να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσει. Όλα αυτά γίνανε στο πρώτο ήμιση του 2011 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εκπρόσωπος των μελών και ένωσης συνεργαστήκαμε εντατικά με Μεξικό, Βραζιλία, με τη ΣΥΠΑ και με ένα σωρό χώρες ε, αφρικανικές στα πλαίσια της ε, οργάνωσης WIPO για να μπορέσουν να προχωρήσει εκεί το θέμα. Πρόκειται επομένως για κάτι το οποίο θα πρέπει να το τονίσουμε. Να το τονίσουμε γιατί έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο κείμενο ε, και να το κατεβάσουμε στην Διαρκή Επιτροπή της που τον Ιούνιο ήδη συνεδρίασε. Με αυτό το κείμενο μπορούμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις και έτσι να μπορούσαμε να προχωρήσουμε χέρι-χέρι με τα κράτη-μέλη για ένα κείμενο λοιπόν το οποίο τώρα ε, έχει λάβει τη μορφή συνετικού εγγράφου όσον αφορά αυτού του περιορισμού, του εθνικού κλπ. Έχει, βρίσκεται επί τη τραπέζη προ τη ζήτηση του ΒΑΙΠΟ. Ε, συζητήθηκε από εμά με Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, ε, Χιλή, Σημερινό, Μεξικό, Νορβηγία, Παραγουάη, Ρωσική Ομοσπονδία και τη ΣΥΠΑ. Οι συζητήσεις από αυτό το κειμένου θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο στην επόμενη συνάντηση στα πλαίσια της ΒΑΙΠΟ και εμείς δε θα, θα συντονιστούμε τα κράτη-μέλη σε σχέση με την θέση που θα αποκρισταλώσουμε. Πάντως ε, στην παρούσα φάση δεν έχουμε αρκετή στήριξη στο Συμβούλιο ούτω ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι αποτελεί συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει το κείμενο που βρίσκεται στους τραπέζε, να το βελτιώσει όσο γίνεται περισσότερο. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούμε και εμείς να εξασφαλίσουμε μια στέρεα βάση. Και αφήσουμε στο μέλλον να πάμε σε συμφωνία. Αυτά. Όσον την Επιτροπή, για το τι έχει μέχρι σήμερα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρο. Νομίζω ότι ε, η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ε, δικαιοσύνη μπορεί να μας πει δύο λόγια σε σχέση με τα θέματα που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Σομελά. Ναι, σας ευχαριστώ στα αγγλικά. Εάν δεν έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, δεν έχω να προσθέσω τίποτα στα όσα είπε από τη Γενική Διεύθυνση Μάρκ, η συνάδελφος. Η πρόεδρο. Καλά, ε, αν χρειαστεί θα λάβετε το λόγο να μα τα πείτε και τώρα. Η κυρία Ντεμπρούν. Σα ευχαριστώ πολύ. Καταρχά ε, με συγκλώνησε η αναφορά του αναφερόμενου σχετικά με την επίσκεψή του στην ε, Δημοτική Βιβλιοθήκη, γιατί εγώ πηγαίνω κάθε εβδομάδα στη βιβλιοθήκη και καθόλου δεν θα μου άρεσε να διαπιστώσω ότι δεν έχω πρόσβαση στο 95% των βιβλίων. Άκουσα με ενδιαφέρον την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διευκρίνησαν ότι το Συμβούλιο τους δίνει την διαπραγματευτική τους θέση. Ωστόσο, αυτό που δεν είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα είναι αν κατά πόσο πλευράς Επιτροπής θα θέλαν να είναι σε θέση να διαπραγματευτούν μια πλήρη συνθήκη και κατά πόσον αυτή η θέση θα ήταν αυτό που θα επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαφώς θεωρώ ότι θα έπρεπε ως Επιτροπή του Κοινοβουλίου να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει την ισχυρότερη δυνατή θέση. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή να το θέσει αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επειδή η Κομισιόν μας λέει ότι το Συμβούλιο διαπραγματεύεται τη θέση που εκπροσωπεί η Επιτροπή, θα έπρεπε ίσως να κάνουμε και μία ερώτηση προς το Συμβούλιο. Επιφυλάσσομαι περαιτέρω σχολείων μέχρι να μας διευκρινίσει η Κομισιόν ποια είναι η θέση της για το ποια θα έπρεπε να είναι η διαπραγματευτική τους θέση, παρά το γεγονός ότι δεν είναι αυτοί που αποφασίζουν. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφος Όκεν. Ναι, καταλαβαίνω ασφαλώς αυτά που είπε η Μπάρμπαρα Ντρεμπρίν, αλλά να προσθέσω ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το Κοινοβούλιο είναι υπέρ μιας δεσμευτικής συνθήκης. Αυτό έχει καταγραφεί αν απλά το ξεχνάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι το, ότι το Κοινοβούλιο δηλαδή συμμετέχει και αυτό στην διαδικασία αυτή, δεν έχει να κάνει μόνο με το Συμβούλιο η διαδικασία αυτή. Όχι, και το, συμβου... και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Να προσθέσω επίσης ότι... ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικυρώσει την ε, σύμβαση των ανάπηρων ατόμων φέτος, όπου στο 30,5 αναφέρεται ότι η νομοθεσία που προστατεύει τα δικαιώματα πραγματικής ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να αποτελεί ένα υπερβολικό φραγμό για τα άτομα με αναπηρίες σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στα έργα του πολιτισμού. Είναι ξεκάθαρη διατύπωση της παραγράφου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ηγείται στις διαπραγματεύσεις για να βοηθήσει τους ανάπηρους για να δώσει υποστήριξη στην αναφορά του Κοινοβουλίου. Αλλά θα ήθελα και εγώ να ακούσω την απάντηση της Κομισιόν πρωτού περάσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ, συνάδελφος Βέρτμαν. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Θα ήθελα μόνο να συμφωνήσω και εγώ με τους δύο συναδέλφους. Αλλά αυτή η εικόνα στη βιβλιοθήκη με άγγιξε πραγματικά γιατί μου αρέσει πολύ να διαβάζω και θεωρώ ότι η παιδεία είναι τα πάντα και ότι η ανάγνωση αποτελεί μια βασική ανθρώπινη ανάγκη και θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Ας φανταστούμε ότι δεν έχουμε πρόσβαση στο 95% των βιβλίων, αλλά ας φανταστούμε ότι αυτό θα αφορούσε δύο άτομα να το πέρα Τι θα κάναμε. Πώς μπορούμε και πώς τολμάμε εμείς να κρίνουμε καν κατά πόσο κάποιον χρειάζεται ένα βιβλίο ή όχι. Γιατί είπατε ότι δεν είναι βιβλία αυτά τα οποία δεν χρειάζονται οι τυφλοί. Μα αυτό πώς να το τολμήσουμε. Σε όλη την λογοτεχνία πρέπει να έχουν πρόσβαση. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν το χρειάζονται αυτό το βιβλίο. Και να σας πω ότι αν θέλουμε θα βρούμε κάποιο τρόπο ακόμα και άτομα με μεγάλες αναπηρίες και αυτό μπορεί να μας αφορά όλους, γιατί ξέρετε όλοι μεγαλώνουμε. Και στην πατρίδα μου έχουμε ε, ένα μέρος όπου ασχολούνται με την ε, φυσική άσκηση των ηλικιωμένων και κάποιος μέτωσε ένα ζευγάρι γυαλιά για να δω πώς βλέπει ένας 80χρονος. Τι να σας πω, επειδή κανείς για παράδειγμα δεν μπορεί να δει καλά, δεν θα πρέπει να διαβάζει. Να σας φέρω τα γελιά αυτά κάποια στιγμή, να δείτε. Πραγματικά αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα. Εγώ λοιπόν θεωρώ προσωπικά ότι πρόκειται για διακριτική μεταχείριση, αν πρόκειται για μειονότητα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Αλλά μιλάμε για διάκριση κατά των ατόμων αυτών σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στα βιβλία στην παιδεία. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ απόλυτη συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το συμφέρον των ενδιαφερόμενων. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Γιάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι προηγούμενοι ομιλητές είπαν τα βασικά και θα ήθελα να εκφράσω την συμφωνία μου Γιατί πολύ απλά δεν ταιριάζει αυτό σε μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία, αν κάποιο τμήμα της κοινωνίας εξαιρείται από την πρόσβαση στην παιδεία και την πρόσβαση στα βιβλία αυτά. Ε, εξαιρούνται, αποκλείεται μια ολόκληρη ομάδα. Αν σωστά κατάλαβα, υπάρχουν πάρα πολλέ συμβάσει, συνθήκε, δηλώσει, πρόθεσει, αλλά αυτό στην πράξη φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Και πάλι έχουμε δύο επίπεδα. Έχουμε το διεθνές επίπεδο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου, απλοϊκά υπομένω. Και αφετέρου έχουμε και την κατάσταση στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν κατανοώ πώς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτουργούν τα πράγματα. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε ως Επιτροπή Έγραψα λοιπόν τέσσερα σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να τονίσουμε. Καταρχάς να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά εκκρεμή. Κατά δεύτερον να υπάρξει σύνδεση με την αρμόδια επιτροπή. Κατά τρίτον θα ήθελα η αναφορά σε οποιοδήποτε μορφή να τύχει διαπραγμάτευση από το Κοινοβούλιο και εξέταση. και κατά τέταρτον θεωρώ ότι μετά τη σύνδεση με την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον ως κοινοβούλιο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το έμεσο δικαίωμα πρωτοβουλίας μας. Καταλαβαίνω τι λέει η Κομισιόν, αλλά το θέμα είναι και η εφαρμογή. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο από τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε την δυνατότητα να ζητήσουμε μέσα δικαίωμα πρωτοβουλίας να ζητήσουμε ε, νομοθετική πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν το θέλει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένη τηλεόγηση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε γιατί προφανώς το ανέφερε με ο αναφερόμενος προς το παρόν η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που θα επιθυμούσαμε. Γι' αυτό λοιπόν Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την αρμόδια επιτροπή. Κατανοώ όμω τον αναφερόμενο. Το αναφέροντα. Πραγματικά είναι κάτι απαράδεκτο για μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία αυτό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι για το θέμα αυτό ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να συγγύσουν και να κάνουν ότι δεν βλέπουν τίποτα. Αυτό το λέω χωρίς οποιαδήποτε διάθεση να προσβάλλω τον οποιοδήποτε, γιατί ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ε, Γενική Διεύθυνση που ασχολούνται με εμπορικά θέματα, ότι πρόκειται για εμπορικό θέμα. Είναι πραγματικά αυτό απίστευτο. Μα εδώ πέρα μιλάμε για ένα ηθικό αδιέξοδο. Τελεία και παύλα. Είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε το δραματικό πρόβλημα εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν έχουν το βασικό δικαίωμα πρόσβασης στο κληροδότημά τους διαβάζοντας πολύ απλά επειδή ένα εμπορικό ζήτημα εμποδίσει τους ανθρώπους αυτούς να έχουν τα βιβλία σε προσβάσιμη μορφή. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό μόνο σε εμπορικό θέμα όταν έχουμε τη δυνατότητα να εξαγάγουμε βιβλία στο σύστημα Braille εκτός Ευρώπης, σε άλλους προορισμούς και παράλληλα αυτά να θεωρήσουμε ότι, α, κοιτάξτε, είναι μόνο εμπορικό το ζήτημα εμπορικής φύσης. Μα όχι, είναι δεοντολογικό το θέμα αυτό και αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό διμερώς πώς θα πρέπει να επιληθεί. Τα κράτη-μέλη με, με τις ε, χώρες εκτός Ένωσης και επίσης ενώπιόν μας μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποια κράτη-μέλη κάνουν ό,τι μπορούν για να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά πάλι όχι. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν με σαφήνεια καταρχάς ότι η αναφορά θα πρέπει να μείνει ανοιχτή. Κατά δεύτερον, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μείνει στην αρχική θέση προκειμένου αυτό να καταστεί δεσμευτική νομοθεσία για όλα τα κρατημέλη και ότι τα βιβλία στο, που είναι τυπωμένα σε σύστημα Braille θα πρέπει να εξάγονται χωρίς τέλη. Και πείτε μας, φίλοι μου, πόσα χρήματα χάνουμε μη επιτρέποντας να τυπωθούν αυτά τα βιβλία σε μπράγι χωρίς πνευματικά δικαιώματα. Φαντάζεστε ότι το δραματικό αυτό πρόβλημα αφορά μόνο για κάποιο περιορισμένο χρωματικό ποσό που χάνουν κάποιοι εκδοτικοί οίκοι και να πούμε ότι εντάξει αυτό το δεχόμαστε και ότι αυτές είναι οι αξίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το αντιμετωπίζουμε σαν εμπόρευμα. Αυτό πραγματικά είναι σοκαριστικό. Και δεν δέχομαι, δεν δέχομαι τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα να μείνει ανοιχτή η αναφορά, προφορικό ερώτημα και ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπογραμμίσουμε την πρόθεσή μας να υπάρξει δεσμευτική νομοθεσία που θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη και έτσι να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξάγει τα βιβλία της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα παραμείνουμε αξιόπιστοι στα μάτια εκείνων που είναι τυφλοί. Τελεία και παύλα και σας ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί έξαφνα στον καθένα μας, να χάσουμε το φως των ματιών μας, λόγω βλάβης, τραυματισμού στα μάτια ή στον εγκέφαλο και να μην μπορούμε να συμμετέχουμε πλέον στην κοινωνική ζωή, γιατί θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο βασικό, θεμελιώδες δικαίωμα, όπως και ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ότι και οι τυφλοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πλήρη λογοτεχνική συλλογή. Αν φανταστούμε για παράδειγμα ότι από αύριο δεν μπορούμε να διαβάσουμε εφημερίδα και βιβλία, θα βρεθούμε στο περιθώριο πλέον της ζωής. Δεν θα ξέρουμε τι θα συζητιέται στην πολιτική ζωή, στην κοινωνία. Όλοι μας είμαστε στην πολιτική. Για φανταστείτε λοιπόν να μην μπορούμε πλέον να συμμετάσχουμε στην πολιτική ζωή. Γι' αυτό λοιπόν και υποστηρίζω την αναφορά και θα ήθελα να αποθύνω έκκληση να, απαιτήσω, να απαιτήσουμε να υπάρξουν δεσμευτική νομοθεσία προκειμένου όλοι οι τυφλοί να έχουν πρόσβαση σε εφημερίδες και στα βιβλία. Και η κυρία Βέρτμαν, ξαναζητάει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και πάλι. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Μποστινάρου και να προχωρήσω και λίγο παρακάτω. Σκεπτόμενοι το εμπόριο και τα προβλήματα σε εισαγωγικά που αντιμετωπίζουν οι εκδοτικοί οίκοι, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι δεν τα πηγαίνουν κι άσχημα οι εκδοτικοί οίκοι και ότι μπορούν να επιδείξουν φιλανθρωπικό έργο και να αποτελέξουν υπόδειγμα στον κόσμο, δημοσιεύοντας αμα, βιβλία σε σύστημα Braille και να κάνει κάποιος την αρχή. Να πει ότι, ορίστε, εμείς δημοσιεύουμε τα βιβλία αυτά. Χωρίς κερδοσκοπικούς σκοπούς. Αν τίποτα άλλο δηλαδή δεν λειτουργήσει, αποτελεί και αυτό μία οδό. Ευχαριστώ, συνάδελφο Αλφάνο. Ε, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ακούγοντα τα όσα είπαν όλοι οι συναδελφοί σχεδόν, αισθάνομαι την ανάγκη να αιτιολογήσουμε το δικαίωμα στον πολιτισμό και στην ε, καλλιέργεια. Ε, ε, κατά τη γνώμη μου ε, δεν συνειδητοποίησαν ε, αυτό που είπαν γιατί ακριβώς το δικαίωμα στον πολιτισμό δεν είναι εμπορικό δικαίωμα. Αν ακούσουμε λοιπόν, αν εμποδίσουμε τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, στην καλλιέργεια, στην εκπαίδευση, περιορίζουμε σε εμά τους ίδιους τη δυνατότητα να επιδείξουμε και να δείξουμε στις επόμενες γενναίες και αυτή τη βασική αρχή σημαίνει πως είμαστε πολύ πίσω. Μάλιστα έχουμε πάει προς τα πίσω αντί προς τα μπρος. Συνάδελφος Όκεν και μετά κλείνουμε όμως. Ε, to put ε, a specific question to Just. Να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Γιατί η Κομισιόν επιμένει στο να αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα μόνο από την άποψη της εσωτερικής αγοράς, ενώ είναι σαφές πως πρόκειται για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για την εξάλληψη των διακρίσεων. Όταν Γιατί δηλαδή να ασχολούμαστε μόνο με τους κακούς ενώ είναι, προ... ενώ είναι ε, θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί ακολουθείτε αυτή τη γραμμή. Σας ευχαριστούμε κυρία Όκεν. Το λόγο έχει η γάμα δέλτα δικαιοσύνη που έλαβε και την ερώτηση και ίσως θέλει κάτι να προσθέσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω πως έχουμε επιμείνει ότι πρόκειται μόνο για θέμα ιστορικής αγοράς. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο κάτι τέτοιο. Δεν το έχουμε πράξει και ούτε πρώτη θέμα θα να το πράξουμε. Ευχαριστώ. Ναι, δεν είναι αρκούσε αυτή η ερώτηση μάλλον. Σημαίνει ότι θα την αναδιατυπώσουμε καταλήλως και θα την υποβάλουμε στην Κομισιόν. Ακόμα μια απάντηση από τη συνάδελφο Ντεμπρούν και μετά θα δώσω το λόγο στον αναφέροντα. Εγώ είχα ρωτήσει κάτι την Κομισιόν, δεν με νοιάζει ποιος θα απαντήσει. Έκανα μια ερώτηση. Τι διαπραγματευτική στάση θεωρεί πως θα πρέπει να έχει η Κομισιόν όταν θα πάει στην WIPO. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την δυνατότητα να διευκρινίσουμε κάποια σημεία τα οποία νομίζω θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε μετά από τις ερωτήσεις των διαφόρων ευρωβουλευτών. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως η Κομισιόν πιστεύει πως οι ενέργειες τις οποίες προβαίνει υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις της για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν έχει γίνει καμιά αναφορά σε εμπορική πολιτική. Έχουμε μόνο απαντήσεις στις ερωτήσεις και στην παρέμβαση του αναφέροντος από την οπτική γωνία που ενδιαφέρει τον αναφέροντα, δηλαδή εξαιρέσεις και περιορισμοί στη copyright. Γι' αυτό το λόγο η απάντηση της Κομισιόν έχει εστιάσει σε αυτό το ζήτημα. Και ως προς αυτό νομίζω πως χρειάζεται να σημειώσουμε τη διαφορά γιατί φαίνεται να μην ήταν αρκετά σαφής ανάμεσα στην κατάσταση εντός της Ένωσης και την κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πιστεύουμε πως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κομισιόν έχει, όπως είπε και η Κομισιόν στην παρέμβασή της, ήδη υπάρχει οδηγία που είναι η οδηγία που έχει σχέση με την εναρμόνιση κάποιων πτυχών του copyright στην κοινωνία της πληροφορίας που προβλέπει τη δυνατότητα ενός περιορισμού για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες συμπεριλαμβανομένων ε, των, όλων των αναπηριών και επίσης όλα τα κρατημέλη έχουν τέτοια δυνατότητα στην νομοθεσία τους. Αυτό που έκανε η Κομισιόν πέρα από την εφαρμογή από πλευρά των κρατών μελών για αυτή την οδηγία είναι η διευκόλυνση των πρακτικών τρόπων που χρειάζονται για την ανταλλαγή βιβλίων σε ειδικό φόρματ. Και αυτό δεν είναι κάτι που αποφασίζει η Κομισιόν, ούτε κάτι που διαχειρίζεται η Κομισιόν. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποια βιβλία ζητώνται από τους τυφλούς, αλλά αυτό που κάναμε είναι να υποστηρίξουμε ένα memorandum of understanding με τη συμμετοχή όλων των συμμετών ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένες και της οργάνωσης που αντιπροσωπεύει ο αναφέροντας για την ανάπτυξη δικτύων εμπίστων διαμεσολαβητών που μπορούν να βοηθήσουν στο να κυκλοφορήσουν αυτά τα βιβλία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αλλά εκείνοι θα πρέπει να δουν ποια είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι ανάγκες του κάθε κράτους μέλους και με τους τους εκδότες θα πρέπει να συμφωνήσουν για την πρόσβαση σε αυτά τα έργα και σε ειδική έντυπη μορφή. Εάν τώρα ρίξω μια ματιά τι γίνεται σε διεθνέ επίπεδο, όπως σας προανέφερα, πρόκειται περί ενός θέματος ε, για το οποίο εμείς προβλέπουμε στις διαπραγματεύση με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των προσδοτήτων μας και εσείς ερωτήσατε τι επιδιώκουμε εμείς όσον αφορά τις επαφές με τον Γάιπο. Εμείς αυτό το οποίο προσδοκούμε επί τη βάση αυτού που πιστεύουμε, δηλαδή νομίζουμε ότι θα πρέπει να καταβληθεί αυτή η σημαντική προσπάθεια για να διευκολύνουμε την ε, διανομή και διάδοση των βιβλίων σε, σε μορφή προσβάσιμη και αυτό χρειάζεται ένα γερό κείμενο και γι' αυτό και όπως εξήγησε ο ε, έχουμε καταβάλει προσπάθεια η οποία προσπάθεια ε, ήταν πιο έντονη το πρώτο ήμιση του ενεστώτος έντος, τόσο ώστε να καταλήξουμε σε το σκήμα, Στο κείμενο αυτό, το οποίο τώρα στις και δεν ευρίσκεται το προηγουμένω και εμείς θεωρήσαμε ότι οι προσπαθειές μας πιάσαν τόπο. Επομένως, μέχρι, τώρα αυτά καταφέραμε και δεν ξέρουμε βέβαια τι μορφή νομική θα λάβει το κείμενο, τι, τι, τύπο θα περιβληθεί αυτό, αυτή η πράξη. Οπότε, αυτό το οποίο χρειάζεται τελικά είναι να υπάρχει μια, σαφήνεια για το κείμενο αυτό και από την άλλη μεριά θέλουμε να ε, έχουν δεσμευτεί οι εμπλεκόμενοι όλοι, να υπάρχει εμπιστοσύνη και έτσι να προχωρήσουμε σε αυτές τις Προς το παρόν αυτά μπορούμε να σας πούμε και βέβαια θα συνεχίσουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε σε εθνές επίπεδο να φτάσουμε στο επίπεδο που έχουμε φτάσει στο στην, στο ιστορικό της Ένωσης. Κυρία Ούκη εγώ θα είμαι σύντομη, διότι ακριβώς, επιβάσκει και όσον εσείς είπατε, θεωρώ ότι όσον αφορά το copyright, εντάξει, αλλά αυτά που είπατε δεν μας καλούν ως προς τα, θεμελιώδη δικαιώματα, δηλαδή μας είπατε τι έγινε και όσον αφορά την Διεθνή Συμφωνία. παρά το ότι υπήρχε υποστήριξη από πλευρά του Αυτό έπρεπε να κάνετε. Και τώρα βλέπω ότι κινείστε από πλευρά copyright και φύγατε από τα ανθρώπινα δικαιώματα και μας λέτε για τους περιορισμούς που υπάρχουν Ελπίζω αυτό να σταματήσει και να αρχίσετε να ασχολείστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε και να προχωρήσουμε προ την έμπληξη του προγράμματο. Και αυτό να αποτελέσει τη βάση των όσων θα κάνουμε. Και γιατί είναι αυτό το οποίο ε, είπατε ότι επιδιώκεται και το είπατε και τι δύο φορέ που λάβετε το λόγο. Η Κομισιόν θα πρέπει να απαντήσει για δύο λεπτά. συγγνώμη, ο αναφέροντα θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνο και θα είμαι σύντομο και δύο. Θα σα αναφέρω πρώτα πρώτα μα είπε η Κομισιόν το διάλογο με του εμπλεκομένου όσον αφορά αυτό το μνημόνιο κατανόηση, το οποίο εδώ πέρα έχουμε προσυγουρεύσει με του εκδότε ε, το 2010 και ε, και εμείς θα έπρεπε να ε, πάυσουμε τη συμμετοχή μας στο διάλογο και αρχίσαμε να κινούμεθα όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις, τις εγκρίσεις με τους ε, εκδότες ε, όπως προβλέπει ο νόμος πνευματικής διοργησίας γιατί είπαμε ότι δεν χρειάζεται αλλού νομοθέτημα όλα αποδίδουν ε, μέσα από το διάλογο και τελικά φτάσουμε στο σημείο να μην έχει μοιραστεί το ένα βιβλίο Επομένω δεν είπα ότι αυτό δεν αξίζει αλλά παρακαλώ καταλάβετε ότι άλλο, άλλο το τι κάνουν οι διαπραγματεύσει και άλλο το κατά πόσο χρειάζεται τα πλαίσια του ΓΑΕΠΑ μια δεσμευτική συνθήκη μας ανέφερε τα της ε, οδηγίας η Κομισιόν, το τι, τι, τι, εξαιρέσεις επιτρέπονται, τι γίνεται στα κρατημέλια, διότι δύο τρίτα των χωρών σε όλο τον κόσμο δεν προβλέπουν παρόμοιες εξαιρέσεις. Η δε συνθήκη την οποία εμείς προτείνουμε θα βοηθούσε να ε, υπάρξουν εξαιρέσεις και σε άλλες χώρες και έτσι να υπάρχει παντού διανοτα διανομής βιβλίων. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε όπως θέλουμε. Και αυτέ οι αδειοτήσει λύνουν κάποια προβλήματα αυτές οι εγκρίσει. αλλά χρειάζεται να υπάρχει το σχετικό θετικό δίκαιο, διότι το δευτερογενέ δίκαιο δεν αρκεί. Σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για το ότι ομόφωνα συμμεριζόμαστε το αίτημα των αναφερόντων και αναγνωρίζουμε την ανάγκη για επιτάχυνση των ε, δραστηριοτήτων για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ολοκληρωμένη νομοθετική αναγνώριση των ε, δικαιωμάτων που δικαίως διεκδικούν. Υπήρξε μάλιστα μια πρόταση να δοθεί στην Κομισιόν η εντολή να προωθήσει αυτή την πρωτοβουλία, την νομοθετική, την Κομισιόν, ε, την Επιτροπή Αναφορών μάλιστα. Μάλιστα από τα όσα είπατε στις παρεμβάσεις ε, θεώρησα ότι μπορούμε να φανταστούμε δύο φάσεις. Πρώτα, μια ερώτηση προς την Κομισιόν για να προσπαθήσουμε να δούμε μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση για τους λόγους που κατά τη γνώμη όλων μας θα έπρεπε να υποστηριχθεί αυτή η υπόθεση από τις ε, βάσεις δικαίου που δεν έχουν αναγνωριστεί εδώ. Δηλαδή περισσότερο είναι θέμα δικαίου παρά ε, οικονομίας ε, και εμπορίου. Να, δώσουμε, να κάνουμε λοιπόν επίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν και έπειτα να αξιολογήσουμε με βάση την απάντηση την ενδεχόμενη ανάγκη υποβολής ε, μάλλον μιας νομοθετικής πρότασης για το θέμα αυτό. Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα κάνουμε μια πρόταση προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης διάταξης, όπου έχουμε διάφορες αναφορές που από κοινού θα εξετάσουμε. Είναι γεγραμμένες στο σημείο 7. Για αυτές τις ε, αναφορές έχω ε, λάβει μια ανακοίνωση για την σειρά των εργασιών. Ευχαριστώ τους αναφέροντες που έβαλαν τάξη στις εργασίες της ε, Επιτροπής μας. Δεν υπάρχουμε και τόσο πολύ χρόνο, γιατί ξέρετε πολύ καλά πως ήδη σας έχουμε ακούσει επανειλημμένος. Πάντως, αν και κατανοούμε την προσπάθεια που καταβάλατε, θα σας ζητήσω να περιορίσετε τις παρεμβάσεις σας, διότι θεωρώ πως σε αυτή τη φάση αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούσουμε την ενημέρωση από της και των αρχών που είναι παρούσες. Διότι νομίζω πως και αυτό είναι το δικό σας ενδιαφέρον ε, παρά να παρουσιάσετε και πάλι τα αίτια ε, της αναφοράς σας που, μπορεί, που βασικά είναι τα ίδια ε, που είχατε παρουσιάσει. Να δώσω το λόγο λοιπόν όπως μου είχατε ζητήσει στον κύριο Πάολο Πριέρη και τον παρακαλώ να μείνει να περιοριστεί στον χρόνο που του έχει δοθεί. Ευχαριστώ.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 Καλημέρα σας κυρίε και κύριοι. Δεν ε, απαντώ στην πρόεδρο Ματζόνη σε αυτά που είπε, αλλά θα προχωρήσω άμεσα στο κείμενο που έχω δώσει και στους Γερμηνείς για να διευκολύνω την εργασία τους. Ευχαριστούμε την πρόεδρο Ματζόνη και όλα τα μέλη της Επιτροπής για, για το ότι μας επέτρεψαν εμάς αναφέροντας της, αναφορά αυτή να υποβάλουμε τίματα σε, ε, σύμφωνα με τα όσα έχουμε υποδείξει ήδη στις αναφορές μας. Κάνουμε μία πρώτη σύνθεση για να να σας παρουσιάσουμε τη θέση μας. Η νέα σιδηροδρομική γραμμή, σχέδιο 6, είναι άχρηστη και καταστροφική. Είναι άχρηστη διότι η Ιταλία και η Γαλλία είναι συνδεδεμένες από μια ιστορική σιδηροδρομική γραμμή που έχει εξυγχρονιστεί πλήρω. Οι εργασίε έχουν ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2010 με επενδύσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας με γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ ώστε να μπορούν να περνούν σειρμοί ε, ε, επιβατικές και, ε, επιβατική και εμπορική. Το 2010 πέρασε μόνο το 1 13 τρίτο της δυνατότητας της ιστορικής αυτής γραμμής, ενώ σπανίως περνούν εμπορεύματα και επιβάτες και δεν προβλέπεται να συμβάλλουν στην οριμότητα των οικονομιών μας. Η κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη έχει περιορίσει τα κιλά που μεταφέρονται σήμερα, ε, απαιτεί ε, δε την ε, βέλτιστη χρήση των εφιστάμενων υποδομών. Μόνο για παράδειγμα να σας πούμε ότι το πρόγραμμα δεν σκοπεύει να, σεβαστεί μόνο ούτε καν το κοινοτικό συμφέρον και είναι καταστροφική για το δημόσια οικονομία της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομίας πόσο θα έχει αρνητική ε, οικονομικό αντίκτυπο. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο και από διεθνεί μελέτε. Το 2003 κάναμε την πρώτη μας αναφορά. Έχουν περάσει σχεδόν 9 χρόνια, αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει στην επιμονή των προωθητών και των εργολάβων που θέλουν να το προωθήσουν και να το υλοποιήσουν προ όφελό του. Η κυβέρνηση τη Ιταλία είναι ε, συνένοχη και συνένοχη με το, τους ε, εργολάβους. Ε, εκατοντάδες ε, καθηγητές ε, πανεπιστημιακοί έχουν υπογράψει σχετική επιστολή που έχουν στείλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ευχόμαστε ότι τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο πλαίσιο του 2014-2020 και το σχετικό πρόγραμμα πλαίσιο να ακυρωθεί αυτό το πρόγραμμα. Ιταλία Μόλις απολέστη ε, η οικονομική στήριξη το 2008, κλήθηκε να δείξει πως είχε ξεκινήσει το εργοτάξιο. Θέλησε να δώσει, να ικανοποιήσει την ε, Κομισιόν και αντί να το κάνει το άνοιγμα της, της, ε, του εργοταξίου, στην ουσία στρατιωτικοποίησε ολόκληρη την περιοχή της κοιλάδας της Σούζας. Είναι ένα μήνυμα υπεροψίας της κυβέρνησης παρά την ε, ειρηνική διαμαρτυρία των κατοίκων της περιοχής. Η Ιταλία δεν έχει καν τους απαραίτητους πόρους στη διάθεσή της. Αυτή τη στιγμή, με τόσο σοβαρή κρίση, σούσες τόσο σοβαρής κρίσης, ε, η απόφαση μιας κυβέρνησης να παταλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ε, μπορεί αυτό να έχει επιρροή στις προσπάθειες της Ιταλίας. Ε, θα πρέπει ωστόσο να διαπιστώσουμε πως οι πληροφορίες που λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την πρόοδο του, προ, του, του, του προγράμματος είναι παραπλανητικές. Να σα δώσουμε το παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν με στο σημείο μάτι τη 7 Σεπτεμβρίου 2011 λέει πω έχουν γίνει μεγάλε διαβουλεύσει με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Κοιλάδα της Σούζα και με τους τοπικούς πληθυσμού και ότι η επιλογή αυτή ήταν αντικείμενο άδικων επιθέσεων από πλευρά των ε, αντιρρησιών. Για την ιδέα αυτή, λέει, τώρα ακολουθούν και οι Ιταλικέ Αρχέ. Τέλο τη παράθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει εδώ πω οι Ιταλικέ Αρχέ έχουν ευθυγραμμιστεί με το αίτημα, λέει, των πληθυσμών. Είναι ψέμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Θέλουμε εδώ να θυμίσουμε πως ε, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των δημάρχων ε, ολόκληρης της κοιλάδας είναι αντίθετες με αυτό το πρόγραμμα. Έχουν γίνει εδώ και χρόνια πολλές διαδηλώσεις όπου συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Να θυμίσουμε ιδιαίτερα εκείνη της 3ης Ιουλίου όπου συμμετείχαν και πολίτες αλληλέγγυοι που προέρχονταν από διάφορες ιταλικές περιοχές και που βία αντιμετωπίστηκε από την αστυνομία και το στρατό. Σας ενημερώνουμε ότι το εργοτάξιο δεν έχει αρχίσει ακόμα. Οι τρέχουσες εσείς αφορούν μόνο την ε, περιχάραξη ενός, ε, ενός ε, οικοπαίδου που, που, όπου κατοικούν, μάλλον που κατοικοεδρεύει αστυνομία και στρατός. Ε, το έχουν, μοιάζει σαν ένα στρατόπεδο εχμαλώτων στο Αφγανιστάν. Καθημερινά Ε, γίνονται σπαταλώνται ένα σωρό ε, χιλιάδες ευρώ λόγω της έλλειψης αυτού του, του, του χώρου. Εμείς έχουμε λοιπόν όχι την εντύπωση αλλά τη βεβαιότητα ότι τα νέα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ιταλία είναι με όλη την ευγένεια που μπορεί να μας διακρίνει αβάσιμα αβάσιμα τα νέα. Σύμφωνα με την Σύμβαση Άρχου, θα πρέπει να δοθεί στου πολίτε ε, μια πραγματική δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη απόφαση. Και όταν αυτή η Επιτροπή ζήτησε τον Οκτώβριο του 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρί να λάβει κατάλληλη απάντηση, ζητήσαμε λοιπόν στη συνέχεια τη συζήτηση που έγινε, η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε να, ε, αποφάσισε να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον μηχανισμό λειτουργία του του τεχνικού παρατηρητηρίου και των, αρχι... και των τοπικών αρχών κτλ. Δεν ε, λάβαμε καμιά απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα αιτήματα που εμεί διατυπώνουμε σήμερα προς την Κομισιόν. Θέλουμε η Επιτροπή Αναφορών, το Ευρωκοινοβούλιο να καταδικάσουν την, τον βίο τρόπο αφαίρεσης ε, της ελευθερία σκέψης και κυκλοφορία ε, των, πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περιοχή που δεν είναι στρατιωτική βάση. Ε, δεν πρόκειται για επαγρύπνηση, αλλά για επίθεση σε όσου ε, πλησιάζουν με. Ε, δακρυγόνα με ε, γκλόμπ και ούτω καθεξής. Θέλουμε να ανεξάρτητη να γίνει η μελέτη για την ε, σκοπιμότητα αυτού του έργου μέσα στο πλαίσιο της Σύμβασης Άρχους. Η Επιτροπή Αναφορών να αναθέσει σε μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων την αξιολόγηση του κόστους ωφέλειας το θέμα του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Η Επιτροπή Αναφορών δεν θα πρέπει να υιοθετήσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρησιμότητα του έργου αυτού υπάρχει σαφή σύγκρουση συμφερόντων και καλούμε να επισκεφτείτε επιγόντως την ε, κοιλάδα της Σούζης και να έρθετε σε επαφή με όλους τους πολίτες, εμπειρογνώμονες, ε, φορείς και οργανώσεις που ε, δρούν πέρα ή κατά αυτού του σχεδίου. Πρέπει να διευρυνθεί η συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Μεταφορών και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμβάλλοντας έτσι στην μελλοντική υλοποίηση όχι του προγράμματος. Έχουμε παρουσιάσει πριν από ένα χρόνο στην ΟΛΑΦ, στον Οργανισμό Καταπολέμησης της Απάτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τρεις καταγγελίες πιθανών απατών για την Ευρωπαϊκή, για κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το πρόγραμμα και δεν έχουμε λάβει ακόμα νέα. Καλούμε λοιπόν την Επιτροπή Αναφορών και το σύνολο του Κοινοβουλίου να εξετάσουν τις καθυστερήσεις σχετικά με τις καταγγελίες μας. Έπειτα, σε σχέση με τον σχηματισμό της κρίσης της Επιτροπής Αναφορών για το θέμα που εξετάζεται σήμερα. Ευχόμεθα αυτά τα έγγραφα να αποτελέσουν τη βάση της έρευνας που θα ξεκινήσει η, Ευρω... Επιτροπή Αναφορών στην Ιταλία. Εμείς εδώ και 22 χρόνια συνεχίζουμε και είναι αναφυσβήτητο ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε με μια τέτοια ε, κατάσταση και ούτε με τις απειλές ούτε με τη στρατικοποίηση της περιοχής θα σταματήσουμε. Η, το κίνημα Νοτάβ είναι εγγύηση για το μέλλον. Περιμένουμε με εμπιστοσύνη τις δικές σας διαβουλεύσεις και σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Grazie. Ε, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πασερότ. Καλησπέρα σας, Πρόεδρε Ματζόνη, μέλη της Επιτροπής Αναφορών, κυρίες και κύριοι. Μετά από ένα χρόνο θα ήθελα να επαναλάβω κάποιες σκέψεις για τη μη σκοπιμότητα της χρηματοδότησης του τμήματος Τεριέσης Διβάτσα, συνδρομικό άξονα Τεριέσης Διβάτσα που έχει ενταχθεί στον άξονα 6. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ακόμα στοιχείο συγκεκριμένο για την αξιολόγηση. Το αρχικό σχέδιο για τη γραμμή Βενετία Βενετία-Τεριέστη που, που παρουσιάστηκε το περασμένο Δεκέμβριο του 2010. Δεν θα παρουσιάσω εναλλακτική μελέτη, αλλά με το πρόγραμμα αυτό που παρουσιάστηκε με κάθε βιασύνη για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα χρήματα, μπορείτε να βρείτε όλες ε, τις ε, αντιρρήσεις που είχαμε προβλέψει πριν από ένα χρόνο. Επιπλέον, το σχέδιο αυτό δεν συνοδεύεται από ανάλυση κόστος ωφέλης όπως απαιτείται από την Ιταλική νομοθεσία. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνοδεύει αυτή την έκθεση θα πρέπει να ξαναγίνει γιατί η γραμμή Βενετία Τεριέστη έχει ε, ε, κατανεμηθεί σε τρία τμήματα. Αυτό δεν προβλέπεται ούτε από την Ιταλική νομοθεσία ούτε από την Ευρωπαϊκή. Μάλιστα, η προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία ε, έγινε δεκτή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας και αυτή η μελέτη θα πρέπει να ξαναγίνει και να ενοποιηθεί. Η περιοχή από τις οποίες περνάει η γραμμή είναι παρουσιάζει πολλές δυσκολίες ε, όσον αφορά την ε, κοιλάδα της ε, Βενετίας υπάρχει πρόβλημα καθίζησης του εδάφους που μπορεί να προκληθεί από την παρουσία διαφόρων ποταμών και καναλιών σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη από υδρολογική, υδρογεολογική και οικολογική μορφή και μάλιστα διέπεται συχνά από πολύ μεγάλες νεροποντές στην περιοχή την ε, σβεστολιθική όπου η γραμμή υποτίθεται ότι θα περνά από διάφορες σύραγγες για πολλές, ε, πολλά χιλιόμετρα υπάρχει πρόβλημα λόγω ποταμών, λιμνών και ε, δεν γίνεται να εντοπιστεί εύκολα η θέση αυτών των σπηλαίων που υπάρχουν παντού σε, αυτά τα, σε αυτή την περιοχή και είναι αναπότρεπτες οι ζημιές στο υδρογεωλογικό περιβάλλον της περιοχής δεν έχουν γίνει κατάλληλε μελέτε ούτε οι με τι τοπικέ αρχέ, και αυτό έχει φέρει πολλέ επικρίσει για το μη σεβασμό αθηνικών και διεθνών αρχών σε σχέση με την ενημέρωση και τη συμμετοχή. Υπάρχει αντίρρηση ε, για διάφορους λόγους στις τοπικές αρχές, ιδιαίτερα στην περιοχή του Βένετο. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες από αυτούς που τους συντάσσει και από αυτούς που τις διαχειρίζεται. Και όσον αφορά ε, τη, τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά. Η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή γιατί μιλάει πολύ γρήγορα και δεν μπορούν οι διερμηνείς να τον ακολουθήσουν. Όσον αφορά τα θέματα μεταφορών, πολύ, σημαντικές, ε, σημαντική είναι η επιβεβίωση από πλευράς ε, του διαχειριστή της Train Italia όσον αφορά τη δυνατότητα της, ε, του σιδηρομονικού δικτύου στην, ε, στο Βένετο, στο Φρίουλι, Λιβενέτσια Τζούλια και στην Σλοβενία. Ε, και παραθέτω υπάρχει πρόβλημα να γεμίζουμε τα τρένα. Αυτό το επιβεβαίωσαν και εκπρόσωποι της RFAE, της Rete Ferroviaria Italiana σε διάφορες θεσμικές επαφές που έχουν καταγραφεί σε DVD το οποίο θα σας δώσω στο τέλος της παρέμβασής μου. Ένας από αυτούς τους υπεύθυνου για την πρόβλεψη και που είναι και, είναι και των πρωτογραμμάτων των Βρυξελών και ε, είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος. Είναι δύσκολο το πώς έγινε, λαμβάνονται υπόψη όλες αυτές οι τεχνικές και οικονομικές πτυχές και πώς περιορίζεται η αιτιολόγηση των, ε, της χρηματοδότησης σε μια πολιτική απόφαση ή όταν πώς κανείς περιορίζεται στο να σεβαστεί τις ίδιες του τις αρμοδιότητες. Υπάρχει ένα, ένας ε, κοινή, μια κοινή σκέψη και βλέπουμε ε, τις, ε, τα προβλήματα και στο Ιταλικό δίκτυο. Αυτές ε, τα προβλήματα μας επιβεώνουν ότι για 10, χιλιά, χιλιόμετρα δαπανήθηκαν 80 εκατομμύρια, 80 δις ευρώ με ένα ποσοστό χρηστών μόνο 5% στο σύνολο των ταξιδιωτών με των σιδηροδρομικών γραμμών στην Ιταλία. Είναι μια πολυτέλεια που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε και δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιου γιατί οι παραδοσιακές μεταφορές που εξυπηρετούν το 95% των ταξιδιωτών γίνονται κυρίως από τρένα ε, τακτικά και αυτά υποβαθμίζεται λόγω της κακής συντήρησης. Καθημερινά γίνονται απεργίες και διαμαρτυρίες για αυτά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε λοιπόν κατασπατάλη στο δημόσιο χρήματος ενώ έχουμε δημόσιο χρέος πάνω από 1980 δις ευρώ. Είναι τρελό να ζητώνται θυσίες από την Ιταλία και να γίνονται διάφορες ε, διάφορες μανούβρες και λιγμοί που πλήττουν ε, την μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού ενώ ε, από την άλλη πλευρά δίνονται χρηματοδοτήσεις σε τέτοιου είδου ε, προγράμματα. Γιατί δεν γίνονται αυστηρές επαληθεύσεις. Όλα αυτά θεωρούμε πως είναι μια τεράστια αντίφαση. Δεν μπορεί να επιτρέπονται τέτοιου είδου χρηματοδοτήσει για επενδύσει που δεν έχουν περιθώριο απόσβεση και που θα δεσμεύσουν για χρόνια την οικονομία ενό έθνους. Η Ιταλική κυβέρνηση και οι ευρωβουλευτέ ε, της Ιταλίας ε, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα ενώ δεν μπορούν να δώσουν τα δικά, ε, δικά τους και το ξέρουν αυτό πολύ καλά αντί να ασχοληθούν με την λειτουργία των υπάρχουσών υποδομών και ενώ ο δημόσιος ε, ε διαχειριστής λέει στις εθνικές γραμμές επενδύστε στην κεντρική Ευρώπη. Ο κύριος Μπριγχόρς το 2010 στην σχετική έκθεση λέει ότι στην Ουγγαρία έγινε δεκτό να βελτιστοποιηθούν οι πάρουσες υποδομές πριν δοθούν χρήματα για νέες ε, δομές για να φτάσουν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για κράτη που έχουν ε, μη ηλεκτροδοτημένες γραμμές με μια μόνο γραμμή. Στη Σλοβενία οι δυσκολίες λόγω των ε, της γεωγραφίας της χώρας και των βουνών είναι τεράστια. Στην ε, Ιταλία τα όρια είναι 160 με 180 χιλιόμετρα την ώρα στα τρένα και ε, η νέα γραμμή αφορά μια πολύ πυκνοκατοικημένη γραμμή. Θα έπρεπε να υπάρχουν ομοιόμορφες παράμετροι αξιολόγησης για να αιτιολογηθούν και να δικαιολογηθούν τέτοιου είδους προγράμματα. Ζητάμε να Μάλλον καλύτερα είναι να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Γι' αυτό και ζητάμε επαλήθευση για τα σημεία που προαναφέραμε, έτσι ώστε να υπάρξει αξιοπιστία ε, και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τέλος, ρωτώ σε ποιο βαθμό η, απο... η δυνατότητα αποδοχής ε, της ε, αναφοράς της κυρίας Πεσότο που υποβλήθηκε το περασμένο Μάιο και με αριθμό 0694 το 2011. Να δούμε τι έγινε και γιατί δεν έγινε αποδεκτή. Μάλιστα δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Πουλό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όσον αφορά την ε, πρώτη αναφορά, Regarding Επαναλαμβάνουμε λοιπόν για την πρώτη περίπτωση Ακριβώ τελούμε να αναμονή αυτών των σημαντικών ανακοινώσεων από πλευρά τη Ιταλική κυβέρνηση και εμεί επομένω πρόκειται να το τοποθετηθούμε. Τώρα, όσον αφορά τον δεύτερο αναφέροντα, ο συνάδελφο ο Τζόναθαν Μπάρκερ θα ήθελα να σα πει για αυτέ τι μελέτε που έχουν αναλυφθεί επίση για να μπορέσουμε να σα βοηθήσουμε σε σχέση με το τι θα κάνουμε όσον αφορά το να καταλήξουν κάπου αυτέ οι προσπάθειε. Θα πρέπει να δούμε τι προβλέπεται στο διάγραμμα 19 Δεκάτου πρόκειται να θεσπίσουμε κάποιες γαθυντήριες για τα δίκτυα και για τη χρηματοδότηση και επίσης υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά ε, το, το Κοινοβουλίο στις 22 και 23 ενδεκάτου η Επιτροπή σας των Μεταφορών πρόκειται να κάνει εδώ μία ακρόαση για τα τα εδώ στο Κοινοβούλιο. Αυτά και τη σκητάλη τώρα στον κύριο Μπάρκερ, τον συνάδελφο για τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω τώρα να απαντήσω όσον αφορά τον δεύτερο αναφέροντα σε σχέση με την περιοχή στεριές της κλπ. Και να δούμε τι γίνεται με αυτό, τη σαλαμοποίηση. Όπως ξέρετε αυτό είναι κάτι μάλλον βασικό για την Ιταλία. Όμως δεν είναι αληθεύει ακριβώς αυτό το οποίο ο διότι στην περίπτωση του Μέστρε και την Ταιριάστη δεν έχουμε σαλαμοποίηση. Έχουμε κατάτμιση των έργων και προγραμμάτων, αλλά όχι σαλαμοποίηση. Σαλαμοποίηση λαμβάνει χώρα. Όταν με ένα συγκεκριμένο τμήμα, α πούμε, στι δομικέ γραμμέ ή άλλου προγράμματο, ε, βγαίνει έξω από την οδηγία η e ΑΕ. Και οπότε τότε ε, δεν ισχύει η οδηγία για κάποια χιλιόμετρα. Όμω εδώ έχουμε τέσσερι διαφορετικέ διαδικασίε e οι οποίε συντρέχουν μεταξύ ε, Μέστρε και τεργέστε. Ε, ένα δεν έχει ξεκινήσει μεταξύ Μέστρη και Ντιβάτσα στην Σλοβενία και επομένως δεν, δεν χωρεί εδώ πριν τη εφαρμογή του, του, αυτού του, του ΙΑΙΕ οπουδήποτε στην γραμμή αυτή. Αυτό ισχύει και επομένω δεν υπάρχει εδώ πέρα περίπτωση παραβιάσεω ε, τη οδηγία. Τώρα επίση για να σα ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο. Ότι έχουμε μια πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2009 η επερχόν 50 που αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει απλώς να κάνουν συμπίλημα πληροφοριών, θα πρέπει να, να, να, να κάνουν επαλήθευση. Θα πρέπει στην Ιταλία υπάρχει μια απόφαση για μια τέτοια μελέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και νομίζω ότι έχουν κινητοποιηθεί οι Ιταλοί για αυτές τι διαφορετικέ διαδικασίες ε, αυτής της ε, μελέτης ε, επιπτώσεων. Τέλος, η σχετική οδηγία αφορά υγεία και περιβάλλον δεν καλύπτει άλλου είδους κοινωνικές επιπτώσεις ή και κοινωνικές. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον αρχιτέκτονα Φεράτσα που αντιπροσωπεύει το Υπουργείο Μεταφορών της Ιταλίας. Εγώ, ευχαριστώ Πρόεδρε, είμαι, αντιπροσωπεύω εδώ το Υπουργείο Μεταφορών και ιδιαίτερα είμαι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων για την Ιταλία. Θα ήθελα σύντομα να απαντήσω στις αναφορές για την γραμμή Τωρίνο Λιών και για την ταιριά στη Διβάτσα και θα ήθελα να μιλήσω για τα βασικά δύο θέματα που εδώ και χρόνια ε, απασχολούν την κυβέρνηση, μάλλον τις διαδοχικές κυβερνήσεις γιατί πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αρχικά Ξεκίνησε τη δεκαετία του 90. Διάφορες κυβερνήσεις λοιπόν ε, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόγραμμα αλλά και άλλα προγράμματα γιατί μιλάμε σήμερα για τη γραμμή των Λιών ως ένα πρόγραμμα ενώ υπάρχουν και άλλα προγράμματα της ίδιας φύσης που αφορούν την επικράτεια της Ιταλίας και τις γειτονικέ χώρες για, τις οποίες, ε, για τα οποία προγράμματα προχωρούν ε, οι εργασίες ε, υπό συνθήκες ασφάλειας και αποδοχής από πλευράς των εν λόγω περιοχών. Όχι μόνο το τρένο ψηλή ταχύτητα, δηλαδή μέσα στην Ιταλική επικράτεια, αλλά και το διασυνοριακό πρόγραμμα σιδηροδρομικής σύνδεσης που συνδέει την Ιταλία με την Αυστρία. Λοιπόν, οι αναφορές αυτές είναι ευρύτατες. Εγώ θα ήθελα να περιορίσω στα δύο κεντρικά θέματα τη δική μου απάντηση. Η υπόθεση της ζημιάς, της καταστροφής. Η γραμμή για την οποία συζητάμε σήμερα, μάλλον στο οποίο αναφέρονται οι αναφορές, δεν είναι πια το πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται. Από το 2005 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολυάριθμες μελέτες και πολυάριθμες αναλύσεις αντικτύπου που τελικά οδήγησαν στην έγκριση ενός νέου αρχικού προγράμματος που εγκρίθηκε από την Διπουργική Επιτροπή για τον Οικονομικό Προγραμματισμό στις 3 Αυγούστου του 2011 Και έτσι προσπαθήσαμε να απαντήσουμε και στις σημερινές αναφορές και πρόκειται κυρίως για ένα πρόγραμμα ε, το οποίο σίγουρα έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις των κατοίκων της κοιλάδας της Ούζε που σίγουρα λόγω ποιότητος και πληρότητος των εκθέσεων προσφέρει εγγυήσεις σε σχέση με τις πτυχές, τις περιβαλλοντικές και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο του προγράμματος. Εμείς θεωρούμε πως αυτό το έργο δεν είναι καταστροφικό, έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Είναι ένα έργο, μάλλον ένα από τα έργα υψηλής ταχύτητας που αποτελούν τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου της Ιταλίας από το 2008 υπήρξε χρηματοδότηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω και χρηματοδοτήθηκαν άλλα 40 ε, ιταλικά έργα. Οι συνθήκε υλοποίηση τη σύραγγα τα μέσα και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ε, πραγματική ανασκαφή είναι οι ίδιες τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την Μητροπολιτική Γραμμή του Τωρίνου, για το μετρό του Τωρίνου δηλαδή, ε, τεχνικές που επέτρεψαν να υλοποιηθεί το μετρό πάντοτε υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και μάλιστα υπήρξαν και, άλλες, ε, και άλλα γεγονότα που οδήγησαν την, το Τωρίνο, την πόλη του Τωρίνο να γεμίσει από τουρίστες. Είχαμε, δηλαδή είχαμε ιδιαίτερα επιβαροντικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Εκεί λοιπόν όπου θα υπάρξει τον, η νέα συνδρομική σύραγγα ε, ήδη γίνεται ότι ανασκαφεί η σύραγγα ε, ενός ε, οδικού, μιας οδικής σύραγγας του Φρεζούς. Είναι μια σύραγγα ασφαλείας που είναι απαραίτητη για να εγγυηθούν με την χρήση των χρηστών της οδικής σύραγγας. Χρησιμοποιούμε τις ίδιες συνθήκες γεωτεχνικές και γεωμορφολογικές. Στο ίδιο βουνό γίνεται αυτή η σύραγγα. Οπότε γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη η σύραγγα η σιδηροδρομική που μάλιστα θα είναι μάλιστα το 88% του ιταλικού κομματιού είναι σε σύραγγα μέσα. Μόνο δύο κομμάτια δεν θα είναι στην ε, σύραγγα, δηλαδή δύο κομμάτια 7 χιλιόμετρων περίπου το ένα θα είναι η σύνδεση με το αεροδρόμιο της Σούζα και το άλλο με το, με αεροδρόμιο του Ορπασάνο. Είναι πολύτιμες περιοχές, ε, όπου πολύ πυκνοκατοικημένες, με σημαντική ανάπτυξη υποδομών. Είναι δηλαδή περιοχές όπου ήδη υπάρχουν ε, μεγάλα οδικά και σιδηροδρομικά έργα. Γιατί είναι απαραίτητη η γραμμή. Λέτε ότι αρκεί η ιστορική γραμμή. Αυτή είναι του 1870-71 η γραμμή και είναι μια γραμμή που αυτή τη στιγμή ε, για λόγους ασφάλειας λειτουργεί σε μία μόνο γραμμή. Μέχρι 1200 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας στάνει υψόμετρο 1200 μέτρα και πρέπει να συχνά χρειάζεται διπλή ή τριπλή μηχανή. Με αυτέ τι συνθήκε η γραμμή αυτή δεν είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι ανταγωνιστική κυρίω με όλε τις άλλε σύραγγε που έχουν φτιαχτεί ε, τα τελευταία χρόνια, σιδηροδρομικέ σύραγγε που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια στι Άλπεις. Να Αναφέρω μόνο τις, δύο σύραγγες που έχει φτιάξει η Ελβετία και που εξυπηρετούν ε, τη σύνδεση Ιταλίας και ε, μάλλον Ελβετίας με Ιταλία κάτω από την Τομοντόσολα και το ιαλι και Άσο Μιλάνο μέσω του σύραγγας ε, Γκοτάρντο είναι απείρως πιο περίπλοκη η κατασκευή τους και ήταν απόλυτη συνένεση των γύρω πληθυσμών. Η ιστορική γραμμή δεν μπορεί πια να λειτουργεί υπό ε, παρά μόνο υπό συνθήκε ασφάλεια, αλλά δεν έχει και τη δυνατότητα πια άλλη ανάπτυξης. Το να σκεφτούμε την ανάπτυξη της ιστορικής γραμμής θα σήμαινε καταδίκη των ενδιαφερομένων περιοχών. Ε, μιλάμε για μια έναν πληθυσμό ε, χρήστες, ε, δηλαδή 17 με 20 εκατομμύρια κόσμο. Δύο κράτη, ε, δύο κράτη σαν το Βέλγιο και την Ολλανδία και που παράγουν 500 δις ΑΕΠ. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε άλλη μια τρύπα στις Άλπεις, ή όχι, αυτό υποτιμά το μέγεθος του έργου αυτού. Ε, θα πρέπει κανείς να σκεφτεί το γεγονός ότι μιλάμε για διασύνδεση ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτά τα έργα εξυπηρετούν τη σύνδεση του Ιταλικού δικτύου με το Ευρωπαϊκό. Δηλαδή θέλουν να ευνοήσουν μια διαδικασία ανάπτυξης στο εσωτερικό ενός προγράμματος και μιας εσωτερικής αγοράς, νέας εσωτερικής αγοράς. Το... Δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη. Πρέπει να υπάρξουν οι ανταλλαγέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γεγονό ότι για αυτές τις γραμμές υπάρχουν αντιρρήσεις εδώ και 20 χρόνια ε, το, το, το έργο έχει αλλάξει πολλές φορές και η θέση μας ε, πάντοτε μιλάει για κάποια βασικά στοιχεία, για τη ζημιά, για τη χρήση, για την, ε, το μεγάλο κόστος αυτής της γραμμής. Εγώ νομίζω πως έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες για να καταλήξουμε σε ένα έργο τελικά το οποίο καθιστά διαχειρίσιμες τις πτυχές που σχετίζονται με το νερό, τον αέρα, και ούτω καθεξής. Πιστεύω πως αυτό το πρόγραμμα, όπως και αυτό του Μπρένερο, αλλά και τις ταιριές της Διβάτσα, είναι καρπή μιας πολύ προσεκτικής αξιολόγησης, στην οποία συμμερίζεται όχι μόνο η Ιταλία, ε, αλλά και η Γαλλία, η Αυστρία και η Σλοβενία και ότι κυρίως Υπάρχει μια λογική μέσα στο πλαίσιο του συστήματος των διευρωπαϊκών δικτύων. Όπως σας είπαμε, τα δίκτυα θα, παρουσιαστούν από τον Αντιπρόεδρο Κάλλα στις 19 Οκτωβρίου και εγώ πιστεύω πως εκείνη την ευκαιρία θα είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ο ρόλος που μπορεί να παίξει το σύστημα των ευρωπαϊκών συστημάτων στην ανάπτυξη της οικονομικής της Ευρώπης, δηλαδή το κάθε εθνικό σύστημα. Και σε αυτή την οικονομική ανάπτυξη να είναι λειτουργική η σιδηροδρομική σύνδεση για να ευνοηθούν οι ελεύθερες συναλλαγές και άρα η διαδικασία ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Υπήρου στο σύνολό της. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, θα μπορούσα και να σταματήσω. Είμαι στη διάθεσή σας φυσικά, ανάλογα με τις ερωτήσεις που θα τεθούν. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον συνάδελφο Wills. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και αναπληρωματική στην Επιτροπή Μεταφορών και πρέπει να πω ότι οι αναφέροντες ε, λένε πράγματα τα οποία μπορώ να επιβεβαιώσω. Ασφαλώς υπάρχει διαφορά για το κατά πόσο νοικοδομείται και κατασκευάζεται μια γραμμή, μια οδός υπερταχεία, όπου πάει κανείς με 180 ή 200 χιλιόμετρα ή κατά πόσον πρόκειται για βελτίωση απλά ε, μιας αρτηρίας. Ε, θα επιβεβαιώσω ότι και οι πολίτες και οι δήμαρχοι έχουν αντιταχθεί κατά του μέτρου αυτού. Με κάλεσαν σε μια εκδήλωση 100 δημάρχων σε ό,τι αφορά την αρτηρία Βενετίας Τριέστης και με πολύ επαγγελματικό και καλό τρόπο μας εξήγησαν ποιες θα είναι οι βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον του έργου αυτού. Μας εξήγησαν ότι ο τουρισμός ε, θα διακυβευόταν στην Βενετία, το πόσμο νερό επίσης αναφέρθηκε ότι πιο πιο σημαντικό θα ήταν να γίνει η σύνδεση με την κυκλοφορία της Βενετίας προκειμένου να μην αναγκάζεται ο κόσμος να πηγαίνει με αυτοκίνητο. Άρα δεν καταλαβαίνουμε απόλυτα. Τώρα που η Ιταλία μας από την οικονομική κρίση, πώς διατίθεται ένα τέτοιο τεράστιο χρηματικό ποσό γιατί ελάχιστα συγχρηματοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τέτοιο ποσό για ένα έργο το οποίο βρίσκει αντίθετη την τοπική κοινωνία. Είναι, Σούζα, είναι πραγματικά έντονη η αντίδραση του κόσμου. Το τούνελ, το φυλάν στρατιωτική. Έγιναν συλλήψεις με πολύ με μη αξιοπρεπείς τρόπους. Το κράτος δικαίου, όπως το γνωρίζω στη Γερμανία, δεν νομίζω ότι εφαρμόζεται πλήρως. Θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν υπάρχει, δεν συνάδει αυτό με όσα θα έπρεπε να υπάρχουν. Και νομίζω ότι καταδεικνύει και το, την αντίσταση του κόσμου. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους κατηγορούμε τους ανθρώπους αυτούς απλά ως εγκληματίες να φτάσει δηλαδή ο στρατός να ε, προστατεύει ένα τέτοιο έργο, θεωρώ ότι αυτό που βρίσκεται είναι πραγματικά ασύλληπτο. Η το Αλπάνο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που δώσατε τη δυνατότητα να επανέλθουν οι αναφέροντες και να εκθέσουν τη θέση τους. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει τίποτα να προσθέσω στα όσα είπανε. Θα ήθελα να στραφώ στην Κομισιόν και στον υπάλληλο του Ιταλικού Υπουργείου ε, Μεταφορών. Νομίζω πως κανείς δεν ε, μίλησε στην ουσία για τα όσα ε, απασχολούν τους αναφερόμενους, τους αναφέροντες. Και εγώ ήδη απόψε θα, ζητήσω από την, θα ρωτήσω την Όλαφ τι γίνεται με τις τρεις καταγγελίες που παρουσιάσατε για να καταλάβω αν τα όσα λέτε είναι βάσιμα, αν θεωρήσαν ότι είναι βάσιμα, αν θεωρήσαν ότι είναι λογικά τα όσα ζητάτε ή αν απλώς αρχιοθετήθηκαν σε κάποιο σιρτάρι. Εγώ δεν ξέρω τι και ποιος, ποιος ενημέρωσε τον πάλο του Ιταλικού Υπουργείου Μεταφορών γιατί λέει το να πει ότι η ιστορική γραμμή του 1860 είναι μια γραμμή που δεν λειτουργεί και που, λειτουργεί μόνο εναλλάξ δεν είναι αλήθεια. Λειτουργεί μια χαρά. Θα πρέπει ωστόσο να πούμε γιατί ίσως θα πρέπει κάποια πράγματα να τα δούμε γιατί δεν, δεν έχετε τη δυνατότητα να το δείτε. Ε, λυπάμαι αλλά τα όσα λέγονται είναι τελείως άλλα ντάλλον. Νομίζω λοιπόν πως θα ήταν ε, σκόπιμο να εστιάσουμε περισσότερο ε, τον ε, στόχο. Η υπάρχουσα γραμμή είναι απαραίτητη και αρκεί. Το γνωρίζουμε ότι το ότι η κυκλοφορία εμπορευμάτων έχει περιοριστεί λόγω της κατάστασης και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμή θα μπορούσαν να έχουν ε, δώσει κάποια καλύτερη δυνατότητα στην υπάρχουσα γραμμή. Να έχει εξυγχρονιστεί κάπως και όταν μιλάμε για κίνδυνο και κανένας δεν μίλησε για κάτι τέτοιο. Μιλήσαμε ανέκαθεν για βία σε αυτή την ε, περιοχή και για αχρηστία, ε, Τη στιγμή αυτή που περνάμε τέτοια κρίση, ιδιαίτερα στη χώρα μας, στην Ιταλία, είναι και αυτή, αυτό το πείσμα το να θέλουν να φτιάξουν ένα έργο που κανείς δεν το θέλει, γιατί εδώ οι πολίτες δεν το θέλουν δεν θέλουν αυτό το έργο. Ασκούν το δικαίωμά τους και έχουν μάλιστα και εκείνοι το δικαίωμα να ζουν εκεί όπου ο καθένας έχει κάνει τις θυσίες του, έχει αγοράσει τα σπίτια του. Έχουν το δικαίωμα να σκέφτονται πως και τα παιδιά τους θα πρέπει να μεγαλώσουν σε μια περιοχή που μέχρι και σήμερα ε, ρηπαίνεται διαρκώς και ε, ε, μολύνεται. Εγώ γνωρίζω τον πληθυσμό της κοιλάδας της Ουζέ. Θα πρέπει να σας πω ότι ντράπηκα πάρα πολύ όταν στατικοποιήθηκε αυτή η περιοχή. Μεγάλη άνθρωποι. Αισθάνθηκε γιατί είναι ειρηνικοί οι άνθρωποι. Όταν πάνε να διαδηλώσουν, πάνε να διαδηλώσουν με... μέσα πολιτισμένα, πολύ πολιτισμένα και κυρίως το κάνουν όλοι ηλικιωμένοι, οικογένειες, παιδιά, γιατί στόχος είναι να υπερασπίσουν ακριβώς αυτά που θέλουν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο μετράνε και κυρίως το χρόνο που βρίσκουν οι υποθετηθέμενες ε, ε, ε, παρεμβάσεις των Black block και των ακραίων ομάδων που πολύ συχνά μπλέκονται και δημιουργούν προβλήματα στις διαδηλώσεις σε διάφορες χώρες. Ακριβώς λοιπόν αυτός όμως είναι ο στόχος, ε, να δεν επιρετεί τίποτα, δεν εξυπηρετεί, δεν έχει καμιά χρησιμότητα αυτή η γραμμή. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα, αφού η Ιταλία μπορεί να τα βάλει αυτά τα λεφτά, αλλά νομίζω πως ούτω ή άλλω η αλλω η ιταλια δεν τα έχει αυτά τα λεφτά και είναι τρελό να ζητάμε τα χρήματα αυτά να τα πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτά που ήδη έχουν δοθεί για να ξαναδούμε και για να δώσουμε μια όθηση στην ιστορική αυτή γραμμή. Πιστεύω πως θα είχαμε ένα αποτέλεσμα εξαιρετικά ισχυρό που θα έχει αφήσει ικανοποιημένου όλους τους πολίτες. Και τέλος, άκουσα πριν από λίγο ότι έγιναν όλες ε, οι έρευνες. Πώς έγιναν αυτές οι έρευνες αφού ακόμα τα εργοτάσια δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. Ή μήπω περιοριζόμαστε περιοριζόμαστε στην περιχαράκωση και μόνο του, της περιοχής. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να συζητήσουμε και είναι σκόπιμο που γίνεται σήμερα αυτή τη συζήτηση να διευρυνθεί για να καταλάβουμε πως δεν είναι κάτι το ακραίο χωρίς ε, αιτιολόγηση και χωρίς αποφασιστικότητα. Είναι μια περιοχή που δεν έχει κανένα λόγο να θέλει να κομματιαστεί μόνο για προσκάρες συμφερέντων ορισμένων. Και τα επιχειρήματα των αναφερόντων ήταν ε, πλήρη, αλλά δεν μπορώ να πω το ίδιο ούτε για την Κομισιόν, ούτε για τους εκπροσώπους της Ιταλικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσω και όλους όσοι μας παρουσίασαν την κατάσταση και μας απάντησαν σήμερα το απόγευμα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα όπου δεν έχω την αίσθηση ότι έχω επαρκείς πληροφορίες στη διάθεσή μου. Καταρχάς το θέμα των τοπικών αρχών και, των... και του κόσμου και τη συμμετοχή του κόσμου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν έχω την αίσθηση ότι έχω μια πλήρη εικόνα και πλήρη απάντηση για το θέμα αυτό και φαίνεται ότι υπάρχουν και αντιφατικές πληροφορίες. Και δεύτερο θέμα, για τον, ε, τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Σημείωσα ότι στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 για την ε, αναφορά του κύριου Παστερούντιου αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μία μόνο μελέτη περιβαλλοντικού ε, αντικτύπου λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα πρέπει να λάβει υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Δεν είναι σαφές από αυτά που μας είπε ο κύριος Πάρκερ σήμερα ότι αυτό είτε έχει ήδη συμβεί είτε πρόκειται να συμβεί. Έλεγε και μιλούσε για κάποιους νέους μηχανισμούς που, έχει, που έχουν καταρτήσει οι Ιταλικές αρχές, αλλά δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε αυτό στην απάντηση των τελικών αρχών. Άρα, δεύτερη ερώτηση είναι μια σαφής ερώτηση και μια σαφής απάντηση για μία ή περισσότερες μελέτες που θα λάβουν υπόψη τις οραυτικές ε, συνέπειες και οι οποίες θα λάβουν όλη τη διάρκεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Όκουν. Ευχαριστώ και εγώ από πλευράς μου για όλες τις παρουσιάσεις. Το θέμα αυτό πραγματικά έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι 7 χρόνια το συζητάμε. Το έχω ακούσει εγώ. Κατά βάση φαίνεται σαν χάσιμο χρήματος. Αλλά αυτό δεν απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει τη σπατάλη χρήματος, να απαγορεύει τέτοια ανόητη συμπεριφορά. Αυτό δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είναι η Ιταλική Δημοκρατία αυτή με την οποία είσαστε αντιμέτωποι. Αλλά Νομίζω ότι θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, γιατί έχουμε ένα νέο κομμάτι, μια νέα πληροφορία. Οι 10 κατευθυντήριες γραμμές και οι κανόνες χρηματοδότησης. Στις 19 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της. Άρα, όποιο και είναι το αποτέλεσμα, καλό θα είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά για να δούμε κατά πόσο θα προσθεθεί κάτι στο θέμα. Ιδάλλως, ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει το έργο αυτό, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε μια ολοκληρωμένη βάση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα τίτεν. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ποστινάρου. Yeah, Δύο μικρές παρατηρήσεις, σύντομε παρατηρήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα είναι προφανές ότι οποιαδήποτε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να συζητηθεί με τι κοινότικέ και τοπικέ αρχέ. Οι πληροφορίε που μόλι λάβαμε μας δείχνουν ότι η συμμετοχή αυτή των τοπικών αρχών και των κοινοτήτων δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Βλέπουμε πάρα πολλές ε, διαμαρτυρίες, ε, βλέπουμε και δημάρχους, φαντάζομαι ε, κάτω είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν κατά το σχέδιο αυτού. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον υπάρχει συμμετοχή, κατά πόσον είναι υπέρ ή αντίθετη σε αυτό το σχέδιο, γιατί δεν υπάρχει και μεγάλο περιθώριο ελιγμών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερη πρόταση, για να το διευκρινίσουμε αυτό, στηρίζω τις ε, ιδέες που εξέφρασαν οι διακεκριμένοι συναδελφοί μου. Άρα και εγώ συμφωνώ να μείνει ανοιχτή αναφορά και να προσπαθήσουμε τις πτυχές αυτές να τις ε, διασαφηνίσουμε στη συνεργασία με τις αρμόδιες Ιταλικές Αρχές και τους αναφέροντες και να καταλήξουμε γιατί αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αν συνέβαιναν τέτοια πράγματα σε μια χώρα που πρόσφατα προσχώρησε στην Ένωση ή στη Ρουμανία, τη χώρα μου για παράδειγμα, θα το καταλάβαινα. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εκεί κανονικά θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί νόμοι. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσει και θα ήθελα <laughs> να ζητήσω από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου αν μπορεί να δώσει τις απαντήσεις που ζητήθηκαν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου, για το κομμάτι των ρινολιών, Η ε, γνωμοδότηση υπάρχει, είναι 760 της 29 η Ιουλίου 2011 και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε και να την ε, δούμε. Το σχέδιο της ε, γραμμής του Ρίνο Λιόνε δεν υποστηρίζεται από, από μελέτη πολιτικού αντίκτυπου. Αυτό ισχύει και για το, ε, τη γραμμή Μέστρε Βενετίας μέχρι Τεριέστη που υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα αλλά όχι για λόγους ε, ε, σκοπιμότητας ούτε για να κρύψουμε τα στοιχεία, αλλά είναι τέσσερα συνδρομικά κομμάτια που είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Και εκεί η αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου για την οποία έκανε λόγος πριν η εκπρόσωπος της ΓΔ περιβάλλοντος γίνεται για τέσσερα κομμάτια, μάλιστα ζωρεύοντας και τον αντίκτυπο των τεσσάρων τμήματων αυτών. Τουλάχιστον θα μπορούσα ε, να διορθώσω αυτό ότι δίθεν δεν έγινε μελέτη του σωρευτικού αντικτύπου. Η ελλειπής τώρα συμμετοχή των τοπικών ε, προσώπων. Δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι δεν έγινε διαβούλευση. Μάλιστα θα ή ότι δεν υπήρξε συμμετοχή και ανάμεξη του πληθυσμού. Υπήρξε και το γνωρίζουμε όλοι για την γνωστή υπόθεση ότι υπήρξε κατασκευάστηκε το παρατηρητήριο τη Κοιλάδα της Σούζα, το τεχνικό, τεχνική διαβούλευση, ήταν ευρύτατες οι διαβουλεύσεις, εν μέρει μάλιστα κάπως ε, καταλάγεσαι και η τοπική αντίσταση έτσι, μέσω αυτή τη δημιουργίας, της διαβούλευσης, αλλά το να λέει κανείς ότι δεν υπήρξε καθόλου διαβούλευση είναι ε, λάθος. Να δώσω ένα λεπτό σε εσά τώρα για να απαντήσετε. Μια διευκρίνηση σημαντική. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος Το Υπουργείο Μεταφορών της Ιταλίας γνωρίζει την υποδοχή της προσφυγής από πλευράς του WWF που μάλιστα κατα... κατένιμε σε τέσσερα τμήματα την μελέτη του περιβαλλοντικού αντικτύπου και την υποδοχή που είχε αυτή η μελέτη και η σχετική προσφυγή. Εγώ έχω ήδη στείλει πριν από κάποιους μήνες ένα αντίγραφο στην Κομισιόν που επιβεβαιώνει αντίγραφο αυτής της προσφυγής που έγινε δεκτή. Ε, είναι λάθος να λέτε λοιπόν ότι είναι δυνατόν να γίνουν τέσσερις ε, μελέτες σε περιβαλλοντικό αντικτύπου χωριστά. Δεύτερη παρατήρηση και λεπτομέρεια. Στις αρχές του έτους έδωσα εγγραφά για το πώς στάλθηκαν τα προγράμματα των έργων στη, στην ε, διοίκηση εντός των προθεσμιών για να υποβληθούν παρατηρήσεις από πλευράς των πολιτών και των ε, θεσμικών οργάνων. Δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες από τον ανάδοχο του έργου και μάλιστα έχω τα πρακτικά για το πότε έλαβαν οι Δήμοι την υποβολή των, των έργων. Και μάλιστα έχω και τα τελευταία, τα τελευταία πρακτικά ενό Δημοτικού Συμβουλίου όπου υπάρχει αντίσταση για αυτό το έργο και προστίθεται αυτό στι αποφάσει διαφόρων άλλων Δήμων. Στην περιοχή του Βένετο κανένα δεν συμφωνεί εκτό από έναν Δήμο για την γραμμή, για την κατασκευή αυτή τη γραμμή. Όλοι οι άλλοι είναι αντίθετοι, κυρίω στο Βένετο. Ε, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε όλα αυτά, κύριε εκπρόσωπε του Υπουργείου. Μεταφορών της Ιταλίας. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ... Ναι, ναι, θα είμαι σύντομος. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια παράξενη κατάσταση. Είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Περιμέναμε να λάβουμε μια απάντηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορισμένοι εδώ κάθονται εδώ πίσω μα και σιωπούν και βάζουν ένα κύριο να μιλάει που από τα λόγια του και από την δύσκολη θέση στην οποία φαίνεται κάλλιστα ότι βρίσκεται, δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά που λέει. Τα λόγια που χρησιμοποιεί ο κύριος Φεράτζα τα, έχουν γράψει άλλοι. Εκείνος απλώ τα διαβάζει ε, και αυτή είναι η αλήθεια. Εμεί λέμε λοιπόν και επιμένουμε ότι όσα λέει ο κύριο Φεράτσα είναι ψέματα. Και μάλιστα μπορούμε να το διατυμπανίσουμε και σα δίνουμε και αυτό εδώ το φάκελο. Ε, σας δίνουμε το φάκελο που λέει τι απαντήσει Είναι εκατοντάδε. χιλιάδες έγγραφα που δίνουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή Αναφορών να σχηματίσει τη δική τη γνώμη. Αλλά εμεί περιμένουμε απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από το Υπουργείο γιατί το να μας δίνει αριθμητικά στοιχεία και, μας δίνει, μας δίνει νούμερα χωρίς να μπορεί να μας τα δικαιολογήσει τα όσα λέει είναι χειραγώγηση. Χειραγώγηση, απόπειρα μάλλον χειραγώγηση τη επιτροπή Αναφορών και των αξιότιμων κυρίων βουλευτών που βρίσκονται εδώ. Μου λυπάμαι που το λέω αυτά αλλά περί αυτού πρόκειται. Σας καλώ Πρόεδρε Ματζόνη να, διαλέ... να διαβάσετε αυτό το φάκελο που σας τον παραδίδω να χείρας για να δείτε ποια είναι η αλήθεια σε αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Σαφώς εμείς ε, λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας και φτιάξαμε αυτήν την ε, ε, αντιπαράθεση, την, ε, μάλλον την κοινή παρουσία σας εδώ. Είναι εδώ η Εκτελεστική Επιτροπή, εκπρόσωποι της Ιταλικής κυβέρνηση, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, όπως έλεγε και η συνάδελφος Άουκεν, εδώ και 7 χρόνια συνεχίζεται αυτή η δουλειά στην Επιτροπή Αναφορών, αλλά υπάρχουν, είναι ακόμα περισσότερα τα χρόνια από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για αυτό το έργο, όπως και για ένα σωρό άλλα έργα που εντάσσονται σε ένα ευρωπαϊκό ε, σχέδιο στο οποίο συμμετείχε η, ευρωπαϊκή, Ιταλική κυβέρνηση διαδοχικές μάλλον ιταλικές κυβερνήσεις και που τελικά εκφράζει μια πολιτική βούληση η οποία οδήγησε στα συμπεράσματα που πιθανότατα θα επιβεβαιωθούν στην συνάντηση της 19ης που επαναλημμένως αναφέρθηκε όπου θα καθοριστούν οι γραμμές ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Τώρα η αρμοδιότητα αυτής εδώ της Επιτροπής είναι να προσπαθήσει να διαμεσολαβήσει ανάμεσα στους πολίτες ε, που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, να προσπαθήσει δηλαδή να λύσει τα προβλήματα. Εμείς κάναμε αυτή τη δουλειά ήδη με την προηγούμενη σύνοδο της Επιτροπής μας που είχαμε βάλει στην ημερήσια διάταξη την αναφορά σα. Επετύχαμε κάποιε ακόμα απαντήσει ε, όσο και αν αυτές δεν ήταν ικανοποιητικέ από την Εκτελεστική Επιτροπή. Σήμερα ακούσαμε και την θέση, την επίσημη της Ιταλικής κυβέρνησης, όσο και αν εσεί δεν την ε, συμμερίζεστε και με μια μοναδική πρόταση ακούσαμε, πιστεύω, από τους συναδέλφους που παρενέβησαν, δηλαδή τη πρόταση του συναδέλφου Μποστινάρο, να ζητήσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις από τις Ιταλικές αρχές. Συμφωνείτε, συνάδελφοι, να ζητήσουμε να διαβιβάσουμε ένα ακόμα αίτημα προς τις Ιταλικές Αρχές, ένα ακόμα αίτημα όπου θα ζητάμε περαιτέρω διευκρινήσεις για τα σημεία τα οποία απαριθμώνται πολύ συγκεκριμένα από τους αναφέροντες όσον αφορά τις ε, παρεμβάσεις τους. Θα ζητήσουμε λοιπόν επικόντως απάντηση και έπειτα θα αξιολογήσουμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Η αναφορά στην οποία για την οποία ρωτήσατε τι συνέχεια δόθηκε στην αναφορά της κυρίας Πεζότο εξετάστηκε από τη γραφείο μας, ε, ευλήθη στην Εκτελεστική Επιτροπή, περιμένουμε απάντηση από εκείνη, αλλά το θέμα, η καταγγελία που περιλαμβάνεται σε αυτή την αναφορά, ε, αφορά το τμήμα Βενετίας Τεργέστης. Ήδη λοιπόν εδώ μερική απάντηση στη σημερινή μας ε, συνάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας ενημερώσουμε για το τι έγινε. Μια ερώτηση και μετά κλείνω. Μιλήσατε για προσφυγή στον Όλαφ και ε, επίσης ε, υποδείξατε ότι στείλατε ντοσιέ Α, περιλαμβάνεται σε το φάκελο που μου δώσατε. Στην Επιτροπή Αναφορών. Εδώ, εδώ, σε αυτό το έγγραφο το έχετε. Μάλιστα, μας το δώσετε σήμερα. Ωραία, λοιπόν. Θα αξιολογήσουμε λοιπόν και αυτό το φάκελο και από αυτού θα σας απαντήσουμε. Κλείνουμε λοιπόν για την ώρα την εξέταση αυτής της αναφοράς. Σας ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ή μάλλον να ζητήσω από τους συναδέλφους στην άδεια να κάνουμε μια αντιστροφή στη σειρά τη ημερήσιας διάταξη ανάμεσα στην 9 και στην 8 γιατί για την δεύτερη είναι παρόν ο αναφέρον, ενώ στην άλλη όχι. Άρα λοιπόν να προσχάρουν ευγένειες απέναντι στον αναφέροντα να αντιστρέψουμε τη σειρά των αναφορών. Δεν υπάρχει αντίρρηση, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Ναυρατήλ για την αναφορά 386 του 2007. Is this working? It is. Buongiorno, Signora Mazzoni. Thank you for the opportunity to address this. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω εδώ για την αναφορά μου αυτή. 386-2007 για την μεταρρύθμιση της ζάχαρης περιέλαβε τον στόχο της βελτίωσης της αντικονιστικότητας, δίνοντας κίνητρα στην αφαίρεση των λιγότερο αποδοτικών εγκαταστάσεων. Αυτό ήταν θεμητό, αλλά δυστυχώς τα πρωτόκολλα και οι μεθοδολογίες που υιοθετήθηκαν δεν ήταν εξίσου αξιοσημείωτα. Η κακή διαχείριση της διαδικασίας της μεταρρύθμισης οδήγησε σε μεγάλη ε, ζημία την Ιρλανδική βιομηχανία και αυτό προκάλεσε την αναφορά μας. Τα ευρήματα του ε, ελεγκτικού συνεδρίου του Νοεμβρίου του 2010 επιβεβαιώνουν αυτά που σας ε, έχω εδώ μπροστά μας στο έγγραφο, ότι υπάρχουν πολλά ελαττώματα και σφάλματα σε ό,τι αφορά και την διαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ε, μη αληθών στοιχείων. Παρακαλώ να δείτε την παράγραφο 24 το Ελληνικό Συνέδριο αποφάσισε ότι δεν υπήρχαν οικονομική δικαιολόγηση για να κλείσει η Ιρλανδική αυτή η βιομηχανία, γιατί ήταν και μία από τα πιο αποδοτικά εργοστάσια στην Ευρώπη. Και η έκθεση υποστηρίζει ότι όχι μόνο υπήρχε κατασπατάληση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αλλά και ότι η Ιρλανδία, χωρίς να υπάρχει λόγος, έχασε μια βιώσιμη βιομηχανία με ευρεία οικονομική και περιφερειακή στήριξη που παρήχε πολλές θέσεις εργασίας. Δύο επαγγελματικέ μελέτες για το μέλλον της ε, παραγωγής σάχαρης στην Ιρλανδία δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2011 που καταδείξαν ότι η επεξεργασία σαχαροκάλαμου αποτελεί βασικό στοιχείο στην ε, Ιρλανδική οικονομία. η εκτιμόμενη τιμή επανακίνησης ενός Ιρλανδικού εργοστασίου επεξεργασίας ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι υπάρχει η εκτίμηση, ότι υπάρχει λόγος που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγήσει το κεφάλαιο αυτό, δεδομένων των προβλημάτων που παρουσίασε η διαδικασία μεταρρύθμισης. Θα ήθελα λοιπόν αντικειμενικά να, να εξετάσουμε τα γεγονότα, ιδιαίτερα την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή Αναφορών να έχει τα εξή υπόψη. Αν το εργοστάσιο ζάχαρη στην Ιρλανδία δεν είχε κλείσει, τα τελευταία πέντε χρόνια θα μπορούσε να έχει ε, κέρδος περίπου 236 εκατομμύρια ευρώ βάσει των ε, προσυμφερμένων τιμών για το ζαχαροκάλαμο και της τιμής αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ζάχαρη. Και το κέρδος αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο. Η Ιρλανδία δεν θα έπρεπε να έχει στερηθεί από μια τέτοια βιομηχανία μεγάλη, ιδιαίτερα στι καιρού τη κρίση που ζούμε, ότι επίση θα ήθελα να λάβετε υπόψη ότι οι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δημοκρατία, τι ίσε οικονομικέ ευκαιρίε και τη δικαιοσύνη. Να λάβετε υπόψη ότι το Ιρλανδικό δημοψήφισμα το 1972 που οδήγησε στην συμμετοχή τη Ιρλανδίας το 1973 στην Ένωση, μεταξύ άλλων βασιζόταν στην ε, ιδέα ότι η ποσόστοση η ετήσια για τη ζάχαρη της Ιρλανδίας ήταν να, έπρεπε να είναι 200.000 τόνοι από μια παραγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο 9 εκατομμυρίων τόνων. Ότι η μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε σε ένα άτομο να περάσει τα συμφέροντά του που λήφθησαν από την Ιρλανδική ποσόστοση χωρίς ε, να υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση. Και αναφέρθηκε ότι το Συμβούλιο δεν είχε προβλέψει ένα τέτοιο μηχανισμό που θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει στα εσωτερικά ενός κράτους μέλους. Και έτσι, σήμερα η ποσόστοση της Ιρλανδίας στη ζάχαρη, η ζάχαρης είναι μηδενική. Επίση η μελέτη καταδεικνύει ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ε, τη χρήση παροχημένων και ασφαλμένων δεδομένων. Όλα αυτά είναι ασφαλώς όχι μόνο λάθος αλλά και νομικώς αμφισβητούμενα. Η μεταρρύθμιση της ζάχαρης ε, υποτίθεται ότι συμπεριέλαβε όλους τους εμπλεκόμενου φορείς. Ωστόσο, σε έξι συνελεύσεις ε, Ιρλανδικής, Ιρλανδικής Εθνοσυνέλευσης, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 2.000 παραγωγοί, κατέστησε σαφές ότι εξετάστηκε μόνο το ενδεχόμενο να κλείσουν οι επιχειρήσεις με ε, αποζημίωση, αποκλείοντας τις τρεις άλλες εναλλακτικές λύσεις της μεθαρρύθμισης και ήταν ε, αποκλειστική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσει ότι ήταν αρκετά σαφείς οι δυνατότητες αυτές θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το να αναθέσουμε σε κάποιον άλλο την αρμοδιότητα για αυτά δεν αναφέρει την ευθύνη του πρωταρχικού φορέα. Οι απαντήσεις της ευρωπαϊκή Επιτροπής σε όλα τα σημεία της ουσίας αποτελούν μάλλον δικαιολογίε και όχι λόγους και η απόπειρα δικαιολόγηση του κλεισίματος του εργοστασίου στο Μάλο είναι πραγματικά απαράδεκτη, δεδομένου το γεγονό ότι το προηγούμενο έτος η ιδιοκτήτρια εταιρεία είχε ξοδέψει 25 εκατομμύρια για τον εξυγχρονισμό του εργοστασίου. Το, μάλλον, το εργοστάσιο του μάλλον δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και να εξεταστεί για κλείσιμο με αποζημίωση. Άρα, Συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω ότι βασιστήκαμε σε εσφαλμένα δεδομένα χωρίς να ζητηθεί η κατάλληλη ανάλυση και χωρίς να συμμετάσχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Άρα, το επίπεδο διακυβέρνησης και διαχείρισης ήταν πολύ χαμηλότερο από αυτό που θα περιμέναμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς ε, η Ιρλανδική βιομηχανία παραγωγής ζάχαρης θα πρέπει να λάβει τις απαραίτητες αποζημιώσεις ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Καταθέτω, κυρία Πρόεδρε, αυτή την ε, αναφορά ενώπιόν σας και στην Επιτροπή σας για την ε, επανόρθωση, αν θέλετε, της Ιρλανδικής βιομηχανίας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την εξέταση της αναφοράς. Ευχαριστεί η Πρόεδρος τον αναφέροντα. Και ο κύριος Φίσερ από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας λαμβάνει το λόγο. Η κυρία Φίσερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι μου προκαλεί ελαφριά έκπληξη το γεγονός, γιατί η αρχική αναφορά του κύριου Ναβατήλ αφορά τη σύσταση μιας ε, βιομηχανίας βιοκαυσίμων στην Ιρλανδία και εκεί, όπως σωστά είπατε, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου α, παραγωγής ζάχαρης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αυτά τα βήματα, αλλά επέλεξε να σταματήσει, να κλείσει το εργοστάσιο του και να λάβει αποζημίωση. Και σύμφωνα με τις ε, πληροφορίες που λάβαμε από την Ιρλανδική κυβέρνηση, πλέον έχει αποχαρακτηριστεί το εργοστάσιο και δεν μπορεί πλέον να αλλάξει, να για να παράγει βιοκαύσιμα. Ωστόσο, κανείς δεν εμποδίζει την οικοδόμηση εργοστασίων βιοκαυσίμων στην Ευρώπη. Είτε με ποσοστώσεις είτε όχι. Σήμερα ο κ. Ναβάτιλ αναφέρθηκε στις ποσοστώσεις παραγωγής ζάχαρης, προφήμων. Άρα και στο σημείο αυτό δεν μπορώ παρά να πω ότι τα αριθμητικά στοιχεία του Ελεκτικού Συνεδρίου αφορούν την μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών ζάχαρης στις διάφορες χώρες και όπως ξέρετε σε μια βιομηχανία όπου η ποσόστοση βρίσκεται στα χέρια 30-40 ατόμων είναι πάρα πολύ δύσκολο να λαμβάνουμε αξιόπιστα στοιχεία για τα περιθώρια κτλ. Γιατί όλα αυτά θεωρούνται και δικαίως απόρριτα των εταιριών. Ακόμα και έτσι όμως τα στοιχεία της μελέτης αντικτύπου μπορεί να μην ήταν τέλεια. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κανείς άλλος α, αυτοί που αποφάσισαν ποια εργοστάσια θα πρέπει να κλείσουν και ποια θα συνεχίσουν. Όχι, οι ιδιοκτήτες των εργοστασίων ήταν εκείνοι που είχαν όλες τις πληροφορίες στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν κατά πόσον θα ήταν βιώσιμο το εκάστοτε εργοστάσιο παραγωγής ζάχαρης μετά από την ε, δημοσίευση των τιμών αναφοράς. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς ε, ασκείται κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δικαίωμα που άσκησαν οι μέτοχοι να δαπανίσουν όπου ήθελαν τα χρήματά τους. Είχε το εργοστάσιο, όπως σας είπα, να αποφασίσει ότι θα κλείσει, να μειώσει την ποσοστοσή του και να παράγει λιγότερο. Δεν επηρέασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόφαση αυτή. Να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι το μέλλον των ποσοστώσεων της ζάχαρης θα αποτελέσει τμήμα της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγροτική πολιτική μετά το 2013 και θα δημοσιευτεί στις 12 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος ζήτησε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Ιρλανδό συνάδελφο κύριο Ναύρατιλ, ο οποίος ε, διεκδικεί αυτά που είπε εξ τη χώρα. χώρας. Πράγματι, είναι εθνικό το ζήτημα, δεν είναι ζήτημα που αφορά ένα εργοστάσιο, μια βιομηχανία. Απλά είναι ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία έχει χάσει μια πολύ επικερδή δραστηριότητα εγχώρια λόγω της ε, πολιτικής που γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής. Έχουμε χάσει πολλά εργοστάσια, πολλές βιομηχανίες λόγω της παγκοσμιοποίησης και δεν μπορούμε να τα ανακτήσουμε. Αν αυτή την βιομηχανία μας να ανακτήσουμε θα είναι πάρα πολύ επικερδής, πάρα πολύ αποδοτική. Και δεν θα χρειαζόμαστε καμία αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγή σαχαρότευτλων στην Ιρλανδία είναι μακροχρόνια, παραδοσιακή. Πολλά ήταν τα εργοστάσια, τέσσερα ε, μάλλον, Κάρλο ήταν δύο από αυτά, ε, ένα μήνα έμεινε στο Μάλλο από τα τέσσερα που είχαμε και παρά τα όσα λέει εκπρόσωπος της Κομισιόν, δεν στο μια εταιρεία να δαπανίσει 25 εκατομμύρια για την αναβάθμιση ενός εργοστασίου ακριβώς ένα χρόνο πρωτού κλείσει. Αυτό θα συνέβαινε αν ε, δεν ήταν η αποζημίωση ε, επαρκής. Το αποτέλεσμα ήταν ουσιαστικά να πάυση να εφίσταται βιομηχανία ζάχαρης. Εμείς θέλουμε να την αναστήσουμε και υπάρχει και αυτή ε, η πρόταση για την ε, παραγωγή βεθανόλης. Ε, δεν θέλουμε να παράγουμε μόνο βεθανόλη. θέλουμε να έχουμε συνδυασμένη παραγωγή. Και όταν υπάρχει το εργοστάσιο θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη δραστηριότητα. Όπως είπε και ο κύριος Ναύρετιλ, υπάρχουν 640 εκατομμύρια ευρώ που δεν έχουν ε, ακόμη γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και 300 εκατομμύρια ευρώ αρκούν για την σύσταση ενός ε, εργοστασίου. Αν έχουμε αυτό το κεφάλαιο, τα υπόλοιπα θα γίνουν από μόνα τους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι συνέβη επίσης ε, στο εργοστάσιο το οποίο αποχαρακτηρίστηκε. Πού βρίσκεται τώρα, στη Ρωσία και στο Ισραήλ. Ω αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Να θα έπρεπε να είναι κάπου στην Ιρλανδία, στο μάλλον ή κάπου αλλού. Επίσης τι προτάσεις για το κεφάλαιο ε, μιλάμε για εναλλακτικέ καλλιέργειε και ο κάθε καλλιεργητής ε, Ζαχαρότευκλου θα σας πει ότι είχε προβλήματα παρά το γεγονός ότι το σαχαρότευλο είναι εξαιρετική καλλιεργία. Όλα αυτά να τα λάβετε υπόψη και ιδίω εν ώψη ε, των εκπομπών του διοξιδίου, εν ώψη τη στρατηγική του 2020, αυτό είναι σημαντικό παράγον. Και επίση έτσι ε, είμαστε μείζονε παραγωγή στην Ιρλανδία και όλα αυτά επομένω ε, κα, κατατείνουν στο να αποτελέσουν κομμάτι αυτή τη στρατηγική του 2020 ένα θέμα το οποίο στο Κοινοβούλιο σα απασχολεί κάθε μέρα. Οπότε, γι' αυτό σας λέω. Πάρα πολύ καλά τα είπε ο Μποσινάρου και εμείς ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δει με καλό μάτι το αίτημά μας διότι θεωρούμε ότι δεν ήταν ορθή η απόφαση στην αρχή και ε, έχουμε άλλωστε και όσα έκρινε το ελληνικό συνέδριο τον Οκτώβριο πέρσι που έκλεισε το εργοστάσιο αυτό είναι ένα γεγονός οπότε ε, αυτός είναι ο, ο μόνος τρόπος να επαναρθώσουμε και να πρετανεύσει και πάλι η δικαιοσύνη, να βοηθήσει το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε η ζαχαροβιομηχανία να μπορεί να ξανασταθεί στα ε, πόδια της και ο μόνος τρόπος είναι αυτός που προτείναμε πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Συνάδελφος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, το ελεγκτικό συνέδριο στην εκθεσή του είπε ότι έχουν τα δίκαια τους οι ετούντες, οι οποίοι ε, τόνισαν το ότι θα πρέπει να γίνει μία αμερόληπτη επαλήθευση αυτών των στοιχείων σε σχέση με όλη αυτή τη χρηματοδότηση που εδώ διακυβεύεται, γιατί επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι στο μέλλον κάθε μεταρρυθμίση της ΚΑΠ όλες οι μεταρρυθμίσεις θα είναι δυνατόν να υλοποιούνται ή θα έχουν κάποιο νόημα. Για κοιτάξτε τι έγινε σε σχέση με την ε, ζάχαρη. Πήγαμε στο 1,2 δις ε, σε σχέση με τα μέτρα. Επίσης, σε αυτό το εργοστάσιο ε, είχαμε το κλείσιμο και είχαμε 3.700 καλλιεργητές και 300 τόσο 340 περίπου που έχασαν τη δουλειά τους και είχαμε επενδύσει 25 εκατομμύριων είχαν γίνει την προηγούμενη χρονιά. Επομένω, κάποιε χώρε όπω και η Ιρλανδία δεν θα πρέπει να δέχονται τέτοια χαστούκια από τι μεταρρυθμίσει και γι' αυτό παρακαλώ ε, να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που κατέβαλαν οι αναφέροντε και ελπίζω ότι θα τίνουμε δίκο σε όσα έχουν πει. Ευχαριστώ. Δεμπρούν. Ναι, και εγώ να προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία ήδη ακούσαμε, ότι δηλαδή πρόκειται για πράγματα τα οποία τα είχαμε πει, τα είχαμε πει με έντονο τρόπο, ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση της παραγωγής και όχι κλείσιμο του εργοστασίου. Και εγώ θυμάμαι ξεκάθαρα ότι η μόνη φωνή που ακουγόταν, η μόνη, τα μόνα στοιχεία τα οποία τότε ήρθανε ήταν ότι η μοναδική επιλογή, η μοναδική λύση, ο μοναδικός δρόμος ήταν το κλείσιμο με παράλληλη αποζημίωση για, για αυτούς θα κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί, γιατί οι κάτοχοι, οι διοκτήτες των ποστόσεων έτσι λέγανε. Δεν ξέρω, αυτά τα ξέρει η Κομισιόν. Τότε πάντως ξεκάθαρα αυτά λέγανε. Σε σχέση με αυτά που εμείς είχαμε προτάξει. Εάν είχαμε δει την άλλη εναλλακτική, τότε θα είχαμε φυσικά και μελέτη αντικτύπων ε, περιβαλλοντικών. Πάντως ομολογώ ότι σαφώς από όσα λένε οι Ιρλανδοί, οι αναφέροντες και οι άλλοι ότι ε, πρόκειται για απόφαση που οπωσδήποτε δεν περιείχε ξεκάθαρα στοιχεία τα οποία εμείς δεν τα ξέραμε. Δεν υπήρχαν δηλαδή όλα τα ορθά δεδομένα σε σχέση με το τι μας εξέθεσε η Κομισιόν, ούτω ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Οπότε διαμορφώθηκε η σχετική πρόταση και έτσι πέρασε και στους υπόλοιπους ο επόμενος. Ναι, εν συντομία να κάνω μια προσθήκη. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα αν ε, είμαστε ειλικρινεί, ε, είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πλέον ε, τον αναφέροντα, γιατί έχει κλείσει το εργοστάσιο και έχει χαθεί η παραγωγή. Αυτό που είναι σαφές είναι το εξής. Δεν είναι δυνατόν να άφησε η Ιρλανδία την παραγωγή ζάχαρης της. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να απευθύνω την εξής έκκληση και να επρασπιστώ κάπως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ποσόστοση για την αγορά ζάχαρης. Ως ε, βουλευτής που ήρθα λίγο αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σας πω ότι είμαι κατά των ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις είτε στο γάλα, είτε στον καπνό, είτε στη ζάχαρη. Σε κάποιο σημείο μας εμποδίζουν στη ζάχαρη είχαμε μια υπερπαραγωγή ζάχαρης κάποια εποχή και με επιδοτούμενες τιμές ε, ασκούσαμε πιέσεις στην ε, παγκόσμια αγορά. Έπρεπε λοιπόν να αντιδράσει η πολιτική αυτό και έκανε. Και μπορούμε να πούμε ότι ήταν επιτυχής αυτή η παρέμβαση γιατί περιορίστηκε η παραγωγή ζάχαρης και ξαφνικά έχουμε το εξή πρόβλημα. Επιβαρύνθηκε η, η παραγωγή ζάχαρης και είναι λίγη πλέον η παραγωγή ζάχαρης στην Ευρώπη. Καλύτερα λοιπόν θα ήταν στα πλαίσια της ε, γεωργικής μεταρρύθμισης να συζητηθεί με την ησυχία μας να συζητήσουμε το θέμα της ζάχαρης, να συζητήσουμε εναλλακτικέ λύσεις και ίσως να έχουμε το θάρρος και την τόλμη να προτείνουμε λύσεις. Είναι τεράστια η αντίσταση στο θέμα των ποσοστώσεων και την κατάρκησή τους ενδεχομένως στο Κοινοβούλιο. Αλλά αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι κάθε περιοχή θα αποφασίζει μόνη της τι σκοπεύει και τι θέλει να κάνει. Κάποια άλλη λύση δεν βλέπω στην παρούσα φάση. Στην παρούσα φάση έχει κλείσει το εργοστάσιο στη χώρα σας. Το μέλλον είναι αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε και μάλιστα με το ολμή και ο συνάδελφος Κέλλη είναι εδώ στην αίθουσα. Θα πρέπει ίσως να τον καλέσουμε στην Επιτροπή για να συζητήσουμε το θέμα της ζάχαρης. Αλλά είπατε ότι παρουσιάστηκαν εναλλακτικές λύσεις σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την αγορά ζάχαρης. Είναι αρκετά έξυπνο αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όρισε ότι δεν θέλουμε να αναστείλουμε και δεν θέλουμε εμεί να αποφασίσουμε πού θα ανασταλεί η παραγωγή ζάχαρη. Αυτό θα το αποφασίσει η κάθε περιοχή. Θα δώσουμε εναλλακτικέ λύσει και θα αποφασίσει. Η χώρα σα ε, επέλεξε να κλείσει ολοκληρωτικά το εργοστάσιο. Εγώ ως ειδικό ε, ως μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, ειλικρινά δεν έχω παρά να σας πω το εξή. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι σήμερα για το θέμα σας. Μόνο το μέλλον μπορούμε να σκεφτούμε. Να δούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Δεν έχουμε άλλους που οποίοι δίνει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Ε, μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατάλαβα τίποτε χωρί να φορέσω τα ακουστικά μου. Ε, πάρα πολλά τα οποία ελέγχθησαν ε, ήταν ορθά και κάποια άλλα όμως ήταν ανακριβή. Και τώρα δεν θέλω να προσβάλλω κανένα όταν λέω ότι δεν ίσχυαν όλα όσα ελέγχθησαν διότι έχουμε αυτή την όλη μεταρρύθμιση η οποία νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ βιαστική έγινε στο γόνατο και εάν θέλετε μαρτυρία περί τούτου πάρα πολλά στοιχεία που κατατίμησε αυτό, διότι είχαμε διάφορες επιλογές ούτως ώστε να υπάρχει κάποιο είδους εισφορά. Αυτή η εισφορά θα δινόταν ε, και θα ήταν ε, όσον αφορά ε, τους, τους, το τον τομέα των εργοστασίων τέσσερις φορές το έσοδα μιας χρονιάς. Επίσης θα είχαμε τη μετατροπή σε εθανόλια. Αυτό θεωρήθηκε το πρόβλημα της οικονομικής ε, πάρα πολύ αμφίβολο γιατί οικονομικά δεν, δεν ήταν δυνατόν να δικαιολογείται το πώς θα γίνουν τα ζαχαροκάλαμα, τα ζαχαρότευτα τέλο πάντων, εθανόλοι ε, και θα φτάνουμε τα, το, το, θα είχαμε τιμή πετρελαίου που πήγαινε στα 150 δολάρια. Ε, το επίσης είχαμε άλλου είδους μετα, μετατροπή, αυτό το οποίο προτάθηκε από εμά και αυτό θα ήταν το πιο σωστό. Τώρα δεν ξέρω ακριβώ ε, τεχνικά πώ γίνεται. Έχουμε, έχουμε σε τρία στάδια προς αυτή τη μετατροπή και στην πρώτη χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλη ε, επεξεργασία τη ζάχαρη και οπότε έτσι ε, έχουμε πάρα πολύ λίγη ζάχαρη που περνάει και αν θέλετε να κάνετε αυτού του είδου την, την κατασκευή προς εθανόλη αυτό είναι πολύ φθηνό. Οπότε, I go back Οπότε και ακολουθήθηκε τελικά αυτό που ακολουθήθηκε, αυτή και είναι η επιλογή. Εγώ όμως θα σας το λέω και θα το λέω για πάντα και το λέω και από την Κομισιόν. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν κανείς να μεταθέτει τις αρμοδιότητες. Μπορεί κανείς να μεταθέτει ε, μόνο ε, όχι την ευθύνη μάλλον, όχι την υπευθυνότητα, αλλά μόνο τις, τις αρμοδιότητες. Και αυτό ήταν βάση ενός πρωτοκόλου. Το έφτιαξε η Κομισιόν και είπε σε κάθε χώρα. Να, αυτοί είναι οι κανόνες, άντε να τους υλοποιήσετε και, ελάτε, και ξανελάτε να μας πείτε τι καταφέρατε. Όμως τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Ιδίω όσον αφορά την Ιρλανδία. Διότι είχαμε αυτό που λέμε ο κελτικό τίγρης. Κάτι δεν την τίποτα για αυτό, στο ότι τώρα ο τίγρης. Ούτε τίγρης υπάρχει, αλλά ούτε και ζαχαροβιομηχανία δεν υπάρχει. Ο δε Κοσμάκης που ήταν εκεί πέρα και ήθελε να κλείσει το εργοστάσιο, ε, αυτοί το θέλανε. Γιατί, Γιατί θέλανε να απελευθερώσουν το, το ακίνητο, το χωράφι και να το εκμεταλλευτούν. Ε, τρομερό λάθος αυτό. Αυτό δεν έπρεπε να επιτραπεί να γίνει. Οπότε, Ποιε ήταν οι βασικέ μεταβλητέ του, του, του, τη παζοκεφαλιά, ότι συμφωνώ με τον κύριο από τη Γερμανία που μα μίλησε προηγουμένω, ότι εάν ήθελε η Κομισιόν ε, έτσι να ρυθμίσει τα πράγματα, τότε αν θέλει να, έχει ποσοστό, οι ποσοστό θα πρέπει να είναι λογικέ. Αν θέλετε να, να διαγράψετε από, τη, από το πρόσωπο τη γη τη ζαχαροβιομηχανία, τότε άντε δώστε 30-40 ευρώ παραπάνω ένα τόνο. Γι' αυτό σας λέω ότι η μεταρρύθμιση ήταν τελείω λάθος και θα πρέπει τα πράγματα να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση. Και η ουσία της αναφοράς αυτή είναι... δώσω το λόγο στον κύριο Κέλ, στον συνάδελφο Κέλλη να κάνει μια πρόταση γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο. Ναι, ναι, πολύ ωραία τα λέτε και ευχαριστούμε, και ευχαριστούμε που δώσατε στο αναφέροντα τη Σκητάλη να, να πει τα θέματα του. Ευχαριστώ και τους άλλους συναδέλφους για όσα είπανε και σας συμπληρώνω ότι θα πρέπει να τα ξαναπούμε, να ξανασυζητήσουμε για το μέλλον της αγροβιομηχανίας στην Ευρώπη, διότι ακριβώς όπως τελικά προέκυψε, αντί να έχουμε επάρκεια, έχουμε ανεπάρκεια. Μόνο 75% είμαστε αυταρχικοί, οπότε θα πρέπει επομένω να κάτσουμε να τα σκεφτούμε τα στην Ευρώπη θα κάνουμε και βεβαίω η Ιρλανδία έχει αποδείξει ότι μπορεί να παραγάγει αποτελεσματικά ε, και δεν είναι θέμα αυτού του, του, του ενός εργοστασίου. Ολόκληρες κοινότητες, ολόκληρες πόλεις, χωριά εξαρτώνται από αυτόν τον κλάδο. Άρα θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η πόρτα, να μείνουν δυνατέ οι δυνατότητε, να τα ξαναδούμε, να επαναφέρουμε την προτέρα κατάσταση και αυτή η ανόητη απόφαση που μα επιβλήθηκε θα πρέπει να ε, αναθεωρηθεί. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Για να συνοψίσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Εγώ από ό,τι κατάλαβα όλοι συμφωνούμε γιατί είναι σκόπιμο να κλείσουμε τη συγκεκριμένο συγκεκριμένη αναφορά, διότι το υπόθεση του αναφέροντα έχει πλέον εξαντληθεί. Αλλά να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα προς συζήτηση, ενδεχομένως εγκαλώντας την Επιτροπή, μάλλον ενημερώνοντας την Επιτροπή Γεωργίας που είναι αρμόδια επί της ουσίας, ώστε να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες ε, για το θέμα. Ε, συνάδελφος Όκεν για αυτό το σημείο. Όποια... Όποια ήταν και η θέση σα για την αγορά τη ζάχαρης, αυτό αποτελεί ένα ελληνικό ζήτημα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε το οτιδήποτε στο μέλλον. Γιατί πολύ απλά δεν έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όχι, είναι εντοιρλανδικό το θέμα. Αυτό δεν το λέω για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Α, απλά θέλω να πω ότι δίνουμε φρούδες ελπίδες στον κόσμο. Ο κύριος Γιάρ. Νομίζω ότι η πρόεδρος της Επιτροπής έχει δίκιο γιατί η Επιτροπή Γεωργίας για την παρούσα φάση θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα της ζάχαρης στην γεωργική μεταρρύθμιση. Θέλουμε να προετοιμάσουμε και μία ακρόαση για το θέμα αυτό στην Επιτροπή. Γιατί στη μεταρρύθμιση της ε, αγοράς ήταν ε, κακές οι τιμές στην αγορά, ήταν μεγάλη η υπερπαραγωγή ζάχαρης. Έχει αλλάξει όμως η κατάσταση. Οι τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι καλές και είναι μάλλον ελπίς η παραγωγή ζάχαρη και αυτό ταιριάζει με αυτά που είπε η Πρόεδρος. Επαναλαμβάνω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχει κλείσει το εργοστάσιο, αλλά υπάρχει και η ζωή μετά. Υπάρχει και το μέλλον και αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε στην Επιτροπή και θεωρώ ότι η Επιτροπή Γεωργίας ασχολείται με το θέμα αυτό. Άρα ήθελα να υποστηρίξω την Πρόεδρο, να πω ότι έχει δίκιο. Επαναρχόμαστε στην ε, πρόταση λοιπόν που διατυπώναμε. Εγώ νομίζω πως είναι εθνικό θέμα, όπου όμως έχει γίνει μέγα άδικο και θα πρέπει να γίνει ευρύτερη συζήτηση. Αν γίνει όμως κάτι τέτοιο, μπορεί το βασικό θέμα να μείνει εκτός. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, το έχει αποδείξει και το ΔΕΚ και άρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως χωριστό ζήτημα μέσα στο κοινικό πλαίσιο, Οπότε αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή του να την κρατήσουμε ανοιχτή. Eh, sul punto, purtroppo, collega Kelly, eh, del fare giustizia. Συνάδελφοι, για αυτό το θέμα της δικαιοσύνης, <clears throat> εμείς δεν είμαστε αυτός ο οργανισμός που θα μπορέσει να προβεί σε ή να εφαρμόσει ε, δικαστικές αποφάσεις. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να καταγράψουμε, να σημειώσουμε, άντε και να διαμεσολαβήσουμε προς τις Ιρλανδικές αρχές με μια επιστολή όπου να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε περαιτέρω τις Ιρλανδικές αρχές για την υπόθεση αυτή και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως ε, το, η αναφορά σε, εδώ σε εμάς θα πρέπει να κλείσει και το θέμα που τίθεται μέσω της αναφοράς μπορεί να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Γεωργίας για τους λόγους που σας ανέφερα. Άρα λοιπόν μπορούμε να στείλουμε ένα γράμμα στις Ιρλανδικές αρχές για να τους ευαισθητοποιήσουμε περαιτέρω και έπειτα να διαβιβάσουμε την ερώτηση στην Επιτροπή Γεωργίας. Οι συνάδελφοι συμφωνούν. Siamo d'accordo. Μάλιστα, συμφωνούμε όλοι. Να σας απαντήσω σύντομα. Ε, πήγαμε στην Κέιπ PMG να μας δώσουν τη συμβουλή τους και ήρθε ένας ανώτερος εκεί, ένα ανώτερος τέλεχος, είδε τι πρόβλεπε το ελληνικό συνέδριο και είπε επιλέξει ότι αυτό εδώ πέρα είναι μαρτυρία μιας ε, τέλειας ανικανότητας, είναι κάτι που πλησιάζει στην, στην παράνοια. Συγγνώμη, συγγνώμη λέει διακόπτη. 97% αυτό, ε, τι να σας πω, έτσι είναι λέει. Ναι, ναι, το κατάλαβα λέει πρόεδρος. Κατάλαβα. Μιλάτε για μια απόφαση για την οποία όμως, επί της οποίας εμείς δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Δεν είμαστε εκτελεστικό όργανο υλοποίησης, επιβολής των αποφάσεων. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως θεσμός στον οποίο προσέφηκε ένας πολίτης, αυτό μπορούμε να κάνουμε να στραφούμε στις Ιρλανδικές αρχές, να τους υπογραμμίσουμε αυτά που μας αναφέρετε και διαβάζετε ε, για να προσπαθήσουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε και να ελπίζουμε ότι θα <laughs> υιοθετήσουν διαφορετική στάση. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να ενεργήσουμε απέναντι στις Ιρλανδικές αρχές. Αυτό είναι, το θέμα. Εμείς φυσικά και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε γιατί τον, θα κλείσουμε την αναφορά. Άμα στείλουμε μια αντιπιστολή, αυτό σημαίνει πως έχουμε ξεκινήσει μια συνομιλία με τις Ιρλανδικές αρχές, πράγμα το οποίο μας ε, καθιστά υπεύθυνο σε θεσμικό επίπεδο. Όμω πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση γιατί δεν έχουμε άλλα επίσημα όργανα μέσα στη διάθεσή μα για να χρησιμοποιήσουμε. Σα ευχαριστώ και περνάμε στο τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση για την αποστολή στην Βουλγαρία. Δεν μπορούμε όμω να το εξετάσουμε το επόμενο θέμα όταν δεν είναι εδώ αναφέρον και δεν είναι εδώ ούτε και εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Γι' αυτό πάω κατευθείαν στο 11 και όχι στο 8 και εδώ το λόγο στην... δίνω το λόγο στην κυρία ε, Όκεν. Ευχαριστώ. Με ρώτησε ο συνάδελφο Ιτρογιάννη κατά πόσο θα μπορούσαμε να τα αναβάλουμε όλα για αύριο και συμφώνησα. Αλλά αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Αλλά εν συντομία, εν συντομία. Νομίζω ότι στην έκθεση αναφέρεται τα όσα συνέβησαν. Μάλιστα. Η έκθεση λοιπόν, το σχέδιο έκθεσης που έλαβα ήταν καλό. Θα ήθελα κάπως να ενισχυθεί η διατύπωση. Γιατί νομίζω ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί σε ό,τι αφορά την περιγραφή. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι σε διάφορες περιστάσεις διοργανώθηκε, διοργανώθηκαν διαδηλώσεις, διοργανώθηκαν με την έγκριση και τη συμμετοχή σε κάποιες περιπτώσεις των αρχών. Γιατί αυτό συνέβη και στην περίπτωση της επίσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά περιστατικά. Ιδιαίτερα αυτό συνέβησαν στην περιοχή Natura 2000. Να καλέσω τους συναδέλφους να υποβάλουν προτάσεις και συστάσεις προτού παρουσιάσουμε την τελική εκδοχή της έκθεσης στην Επιτροπή. Και πολύ λυπάμαι που δεν το έκανα αυτό προηγουμένως. Είχαμε και πολλά στην Δανία να κάνουμε τον τελευταίο καιρό και σας δώσω συγγνώμη. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να με βοηθήσετε στην συνέχεια της δουλειάς αυτής. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη και θα πρέπει να τονίσουμε την δύσκολη κατάσταση στην περιοχή. Το μόνο που μπορώ να πω για την έκθεση αυτή είναι ότι είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά ίσω δεν αποτυπώνει αυτά που είδαμε ακριβώ. στην ίδια έκταση. Δεν είναι Μποστινάρο. Ευχαριστώ. Άλλο θέλει το λόγο ο κύριο Μποστινάρο. Ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω ιδιαίτερος την εισηγήτρια για το έργο που επιτέλεσε η κυρία Άουκεν η έκθεση εκφράζει ακριβώς τα όσα διαπιστώσαμε στη χώρα και πάλι να ευχαριστούμε την κυρία Αντέλτσεβα και τους άλλους βουλγάρους συναδέλφους που μας ακολούθησαν, μας συνόδευσαν σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης στη Βουλγαρία. Επίσης συμφωνώ με το όσο είπε η κυρία Ούκεν, ότι κάποια συμβάντα, ας τα πούμε, όπως ε, ε κάποιες διαδηλώσεις, κάποιες εκδηλώσεις αυθόρμητες αλλά πολύ καλά οργανωμένες για, για, το πρόγραμμα ε, θα πρέπει να αποφεύγονται στο μέλλον. Πάση θυσία, διότι θυμίζουν την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτά δεν πρέπει να επανελθούν ποτέ. Δεύτερον, θέλω να σας τονίσω ότι τότε που πήγαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ε, ήταν πάρα πολύ θετική η εντύπωση από την Υπουργό, όμως η εφαρμογή των όσων είπε σε τοπικό επίπεδο η εφαρμογή ε, υπολείπεται του, του επιθυμητού υπάρχει κάτι σαν κενό, χάσμα μεταξύ της κεντρικής εξουσίας και των τοπικών αρχών. Οπότε, ό,τι τυχόν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβλάτη μπορεί να συμβεί με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι αντιβάνησε σε νόμους και κανόνες, εθνικούς, ε, ε λοιπά Και ξέρετε αυτά όλα τα ξέρω από τη δική μου χώρα. Α, ρίχτε μια ματιά και στι αναφορέ που θα συζητήσουμε αύριο που αφορούν τη Ρουμανία. Άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό το θέμα αυτό, πάρα πολύ σημαντικό για την Κομισιόν, για τη δική μας Επιτροπή και γι' αυτό και τώρα θα πρέπει να κάτσουμε για να δούμε το πόσο λίγα στοιχεία μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε από κοντά τις ε, εξελίξεις στη Βουλγαρία. Και πού στο, στο ε, σε εκείνη τη χωματερή. Συνεχίζεται βέβαια εκεί η προσπάθεια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πρώτα-πρώτα πώς γίνεται η εφαρμογή των όσων προγραμματίζονται. Πώς εμπλέκεται η κοινότητα σε έναν θεσμικό χαρακτήρα διάλογο με τις ε, αρχές που αυτό πρέπει να είναι υποφελία και των δημοτικών αρχών και του, των, των κατοίκων. Επίσης υπάρχει τώρα και κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά τα, τα, όρια της Ρίλα ότι εδώ έχουμε διαφορετικά επίπεδα συνομιλητών. Εντάξει, όλα καλά. Αλλά εκεί στα βουνά ήταν το αντίθετο. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω Καμιά φορά θα πρέπει ο Επίτροπος να καταλείπει το γραφείο του και να πηγαίνει και επιτόπου για να κοιτάει τι γίνεται, τι γίνεται επί Όταν έχουμε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις που εδώ φωτίζονται εδώ ενώπιον της Επιτροπής μας. Γιατί μιλάμε για εκατοντάδες ε, αναφερόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι προσφεύγουν και θα πρέπει να καλύπτονται. άλλος. Ιδάλλως να συνεχίσουμε να ικανοποιούμεθα από όλα αυτά τα στρογγυλά που μας λέει το Βουκουρέστι, η Σόφια, δεν ξέρω ποιο στην Ευρώπη, αλλά άλλο τα λόγια και άλλο πραγματικότητα που είναι συνήθως αντίθετη. Επίσης να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους της συναδέλφου Γιώτοβα, η οποία και εκείνη ε, συμμετέσχε στην αντιπροσωπεία, ε, ευχαριστεί διότι αναδείχθηκε το θέμα στη Βουλγαρία. Αναδείχθηκε το πρόβλημα το περιβαλλοντικό. Λοιπόν το θα πρέπει να τονιστεί το, το ότι οι αρχέ πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρά τι περιπτώσει αυτέ, τα προβλήματα αυτά και θα πρέπει η, η περίπτωση αυτή τη χωματερή του σχοντόλου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υποφελία ε, και του λαού και του κράτου. Πολύ αξιολογή η έκθεση, η ισόρροπη, όπως η Μαργαρίτα Όκεν μας την τίμασε με Δεν μεταφράζεται. Αγγλικά. Πάρα πολύ καλή έκθεση, λέει κύριε Ναντέλτζεβα. Καλύπτει πάρα πολλά θέματα αυτή η έκθεση και βασίζεται σε κάποια μερόληπτα στοιχεία, όπως το επιτόπου διαπιστώσαμε ότι έχουν και ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συνάντησαν τους αναφέροντες. Τώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια θέματα και έχω και κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά τις ε, διευκρινήσεις, Μιλούμε για αυτούς τους ε, αναφέροντες που αφορούν αυτό το τελεφερίκ. Μιλάμε για 30.000 ε, άτομα μόνο τον Αύγουστο. Ε, είπαμε ότι έτσι έχουμε μειώσει τα προβλήματα της συγκοινωνίας, αλλά έστω και αυτές οι λίγες πληροφορίες που έχουμε βοηθούν έστω και για αυτή την τουριστική περίοδο. Τώρα όσον αφορά τις συστάσεις της, της, της έκθεσης, λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για να έχουμε κάποιο είδους ε, διαρθωτικά προγράμματα και σας υπενθυμίζω ότι οι κατευθυντήριες γραμμές ήδη προβλέπονται, ήδη υπάρχουν και ήδη ε, ακολουθούνται. Όμως έχουμε εδώ δύο συστάσεις πάρα πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε κύριε Όκεν γιατί είναι αλήθεια ότι η απάντηση για όλες τις αναφορές βγαίνει μέσα από το διάλογο με τις αρχές και με τις κοινότητες. Επομένως θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία ε, όλες οι πλευρές και επομένως έτσι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα όπως διαπιστώσαμε ότι ισχύει τόπου στη Βουλγαρία. Ε, επίσης υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία για διεξαγωγή διαλόγου με τις αρχές, όμως από την άλλη μεριά οι τοπικές αρχές πολλές φορές ε, δεν επιδιώκουν το διάλογο, προτιμούν να παραπέμψουν, να προτιμούν το, τα θέματα όλα να ρυθμιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, ε, νομίζω ότι η συστάση και Σάκη είναι πάρα πολύ εύστοχες, να ευχαριστούμε, διότι έτσι είναι εδώ να επιτευχθεί η λύση πώς μέσα από τον διάλογο ε, και έτσι να χρησιμοποιηθεί με τρόπο αποτελεσματικό και από τους διαχειριστές του έργου και από τις αρχές. Και γι' αυτό ε, είναι σωστό αυτό που λέγεται ότι θα πρέπει η Κομισιόν να παρακολουθήσει την, την εξέλιξη σχετικά με κάποιες ε, αναφορές. Όμως θα ήταν πιο σωστό εάν η, δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή Αναφορών, να εστιάσει την προσοχή της σε κάποιες συγκεκριμένες αναφορές, ούτως ώστε οι Βούλγαροι πολίτες να μην ε, θεωρήσουν ότι υπάρχουν ε, αναφορές πρώτης και άλλες που είναι β' κατηγορίας. Επομένω, πάρα πολλέ αναφορέ ε, είναι πάρα δυνατόν να τι εκμεταλλευτεί κάποιο για πολιτικού λόγου. Εμεί όμω, ω Επιτροπή των Αναφορών, δεν θα πρέπει να παίζουμε σε αυτή την παγίδα. Επομένω, εμεί, η Επιτροπή των Αναφορών, θα πρέπει να διατυπώσουμε κάποιε συστάσει. Θα πρέπει να προτείνουμε η δική μα Επιτροπή να παρακολουθήσει την ε, υλοποίηση των όσων συστήνονται για αυτέ τι αναφορέ ε, για τις συστάσεις που απαραίουν από αυτή την αναφορά. Γι' αυτό ε, και πάλι σας ε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι κατάφερε η Επιτροπή των Αναφορών να αποφύγει την πολιτική εκμετάλλευση του θέματος. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους. Ήταν πάρα πολύ επαγγελματικός ο τρόπος που ε, ρυθμίσατε το θέμα και πάρα πολύ ευχάριστη συνεργασία. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εν συντομία και θα ήθελα να σας ε, καλέσω να καταθέσετε τροπολογίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με τις αναφορές. Κάτι άλλο που ανακάλυψα πρόσφατα, για παράδειγμα. Και φοβάμαι όταν κοιτάξαμε και περάσαμε το αιωλικό πάρκο έχω την αίσθηση και λυπάμαι που το λέω ότι μία από τις πρεσβείες, ε, ίσως και η Δανέζικη, έχει κάνει λόμπι εκ μέρους της βιομηχανίας προκειμένου οι αρχές να υποβιβάσουν και όχι να αναβαθμίσουν την περιοχή. Τα κοιτάω αυτά τα θέματα γιατί εξέτασα και περιπτώσεις στην Πολωνία και το διαπίστωσα σε πολλές χώρες ότι οι πρεσβείες μπορούν να αγοράσουν βοήθεια από τα λόμπι. Άλλο να ανοίξουμε πόρτες για νέες βιομηχανίες και άλλο να κάνουν λόμπι, γιατί έτσι κάνουν κατάχρηση της τάσης που έχουν σε μια χώρα. Και είδαμε πρόσφατα με εμπλοκή της Δανέζικης, της Βρετανικής και Γερμανικής πρεσβείας και της Γαλλικής πρεσβείας τέτοια περιστατικά. Θα πρέπει λοιπόν να ανακαλύψουμε τι κρύβεται από πίσω και εμένα μου δόθηκε η εντύπωση ότι το ίδιο ισχύει και για την Βουλγαρία. Φυσικά αυτό δεν μπορώ να το αναφέρω στην έκθεση φέτος, αλλά θα πρέπει να ερευνήσουν τα θέματα αυτά και να δούμε σε πόσες περιπτώσεις οι πρεσβείες χρησιμοποιούνται ως εργαλεία της βιομηχανίας, του βιομηχανικού κλάδου. Επιπληρωμή Τροπολογίες λοιπόν για να ενισχύσουμε την διατύπωση γιατί η κατάσταση είναι χειρότερη από αυτή που φαίνεται στην έκθεση. Ευχαριστούμε συνάδελφε Όκεν. Ήταν μια πρώτη ε, παρουσίαση. Μετά θα υπάρξουν οι προθεσμίες για την υποβολή των τροπολογιών. Θα συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι έτσι και θετικά δεχόμαστε την ε, πρόταση και του συναδέλφου Μποστινάρου να δίνουμε όλο ένα και περισσότερο σε αυτήν την ε, ε, τροπολογία, σε αυτή την μάλλον την Επιτροπή, να μπορέσουμε να ε, σταθούμε στο ύψος μας, να μην πάμε εκεί για να ζητήσουμε το χειροκρότημα της αίθουσας, αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει επί τόπου. Σας ευχαριστώ τέλος των εργασιών της Επιτροπής και αν μου το επιτρέπετε ε, να κλείσουμε αμέσως και να αρχίσουμε την συνεδρία των συντονιστών.